Καλησπέρα. μέρα. Καλημέρα σε όλους και όλους. Ας υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. Βλέπω δεν έχουμε και πολλούς παρόντες, αλλά ας ξεκινήσουμε γιατί θα μας επισκεφθεί σήμερα η Επίτροπος Μάλστρομ στις 12.30 στην συνάντηση των συντονιστών. Οπότε θα πρέπει μέχρι τότε να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το χρόνο μας. We can discuss all of the points θα πρέπει να έχουμε μέχρι τότε ολοκληρώσει όλα τα σημεία της ημερησία διάταξη. Λοιπόν, καταρχήν υιοθετούμε την ημερησία διάταξη με την ακόλουθη αλλαγή. Σημεία 9 και 10 ε, θα τα χειριστεί ε, από τις 12.30 μέχρι τη 1 ε, η πίτροπος Μάλστρομ ε, εκτός της, του συνήθους χρόνου συνεδρίασής μας. Ε, θα συζητηθεί το θέμα των καταστάσεων ε, επιβατών με τους ε, ε εισηγητές, με τον εισηγητή και τους και εισηγητές μόνον. στη μία η ώρα το μεσημέρι, η διαπραγματεύτρια της Επιτροπής, η κυρία Λεμπάγη, διαπραγματεύτρια τη Κομισιόν για το θέμα τη ε, Συμφωνία Προστασία Δεδομένων Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ θα ενημερώσει του συντονιστέ, τον εισηγητή και του σκιώδει εισηγητέ ε, για το στάδιο των εργασιών ε, στη διαπραγμάτευση αυτή τη συμφωνία. Όπω σα είπα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το χρόνο μας γιατί η κυρία Επίτροπος, η κυρία Μάλστρομ ε, θα πρέπει να συμμετάσχει στη συνήθη ε, συνάντηση των Επιτρόπων του, της Ομλέρης Επιτροπής ε, που γίνεται τις Τετάρτες. Από τις 6.30 μέχρι τις 7 θα συναντηθούν οι συντονιστές. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, υιοθετούμε έτσι την ημερησία διάταξη. Και περνάμε σε ανακοινώσεις του Προέδρου. Ε, θα ήθελα να εγκρίνουμε τη σύσταση των συντονιστών για το διορισμό των, εξα... των ακόλουθων εισηγητών. Την κυρία Μποσκούρτ ως εισηγήτρια για την ε, ανάπτυξη ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού. Η Επιτροπή Κάλτη είναι η ε, κύρια Επιτροπή. Μετά, το διοσμό της κυρίας Γκέπχαρτ ως εισηγήτρια για την νομοδότηση επί αποφάσεων σε θέματα ε, οικογενειακού δικαίου. Και επίσης υιοθετούμε τα πρακτικά, σημείο 3 σε τα πρακτικά της συνεδρίας της 21ης και 22ης Ιουνίου. Σας ανακοινώνω επίσης ότι θα λάβει χώρα μια συνάντηση των ε, συγγνώμη. Σας ανακοινώνω ότι θα λάβει η χώρα μια συνεδρία στις 21 και 22 Ιουνίου. Περνάμε στο σημείο 4 της η έκθεση σχετικά με την πρόοδο του κοινού στα έγγραφα. Έκθεση Χαουτάλα. Είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο διότι εξετάζει την εφαρμογή του κανονισμού ως εργαλείο του πολίτη για να ελέγχει και να έχει πρόσβαση στις εργασίες των γραφείων και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ταυτόχρονα εξετάζει θέματα που έχουν σχέση με την ε, πρόσβαση των εγγράφων, διοργανικά θέματα σε σχέση με την πρόσβαση των εγγράφων. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 30 Μαΐου στις 12 ε, το μεσημέρι, ενώ η ψηφοφορία θα γίνει στις 15 Ιουνίου. Ο λόγος στην κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που επανερχόμαστε, που επανέρχομαι στο θέμα αυτό που είχα ήδη ξεκινήσει παλιότερα με τον κύριο Κάσμαν. Ο κύριος Κάσμαν είναι ο εισηγητής για την αναδιατύπωση της οδηγίας στην ε, δημόσια πρόσβαση, ενώ εγώ ασχολούμαι πιο πολύ με την εφαρμογή και τις καινούριες απαιτήσει που προκύπτουν από τη συνθήκη της Αβώνας. Ε, επέλεξα την εξή μέθοδο. Μίλησα με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά χρησιμοποιούν και αποφελούνται αυτού του κανονισμού. μέσω αιτημάτων προς τα όργανα ε, και ε, επανέρχονται αν, ε, με καινούριες αιτήσει αν ε, απορριφθεί πρώτη τους αίτηση ή προσφεύγουν ακόμα και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ο οποίος πραγματικά έχει τα τελευταία χρόνια υποστηρίξει πολύ τέτοιου είδους διαδικασίες. Η το πρώτο τμήμα της έκθεσής μου αφορά τις ε, αλλαγές στο πρωτογενές δίκαιο. Την συνέχιση της με άλλα λόγια, που καθιστά την πρόσβαση στα έγγραφα ε, δικαίωμα του πολίτη, ε, δεσμευτικό δικαίωμα. Ε, θα πρέπει όλες οι αποφάσεις που αρνούνται τέτοιου προσβάσεις να βασίζονται σε πολύ συγκεκριμένους και απτούς λόγους καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει μοντέλο για διαφάνεια και για συμμετοχή δημοκρατία. Ε, η συνθήκη Λισαβόνας ε, απαιτεί επίσης ε, να δίδεται πρόσβαση και σε έγγραφα άλλων οργάνων, όχι μόνο των τριών βασικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει αυτοί οι κανόνες να αρχίσουν να εφαρμόζονται και να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό για την δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα. Ως ε, πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το πώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα εφαρμόσει αυτούς τους κανόνες, γιατί πιστεύω πως ε, έχει έρθει η στιγμή και η εξωτερική μας πολιτική να είναι ανοιχτή στους πολίτες, βέβαια με συγκεκριμένους περιορισμένους ε, περιορισμούς. Ε, δεν ε, μπορεί όμως η εξωτερική πολιτική να ε, είναι προσβάσιμη <laughs> μόνο στους διπλωμάτες και τους πολιτικούς. Η νομολογία έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν απόλυτα δικαιώματα βέτο για την πρόσβαση σε έγγραφα που προέρχονται από τα ίδια. Γιατί ακόμα και όταν αυτά τα έγγραφα έχουν, προκύπτουν από ε, τα κράτη-μέλη τα οποία τα έχουν διαβεβάσει σε όργανα της Ευρωπαϊκής ε, η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους ίδιους κανόνες. Ε, επίσης υπάρχει και ένα θέμα, υπάρχει το εξής θέμα. Τα όργανα πολύ συχνά προστατεύουν προνόμια διαβαθμίζοντας ή υπερβολικά πολλά έγγραφα ή υπερβολικά μεγάλα κομμάτια εγγράφων. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εφαρμογής εκεί πέρα, γι' αυτό το λόγο ζητώ ε, να ρυθμιστεί. Ε, μάλλον ε, ζητώ ένα καινούριο κανονισμό ή τη συμπερίληψη όλων των εγγράφων των οργάνων σε αυτόν τον κανονισμό. Ο κ. Κάσμαν θα ήθελε να δει όλους τους κανόνες διαβάθμισης σε αυτόν τον κανονισμό, εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ ότι ένας διαφορετικός κανονισμός θα περιελάμβανε τους κανόνες διαβάθμισης των εγγράφων, ε, ξεχωριστός κανονισμός ο οποίος θα μπορούσε ε, να υιοθετηθεί κάποια στιγμή. Μετά το πώς εφαρμόζουν τα όργανα τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο κανονισμός στο άρθρο 4 οι βασικές μου παρατηρήσεις είναι οι εξής. Πρέπει να βρούμε μια καινούργια διατύπωση ε, για το, την έννοια του χρόνου προβληματισμού. Ε, θα πρέπει δηλαδή να δίδεται ε, κάποιος χρόνος στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σκεφτούν το θέμα πριν δώσουν πρόσβαση. Όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί αν για παράδειγμα επιλέξουμε να αλλάξουμε τον ορισμό του εγγράφου, τότε ε, θα, θα μπορούσε να διευρυνθεί πάρα πολύ το πεδίο αυτής, ε, αυτού του χρόνου προβληματισμού. Ε, νομίζω ότι αυτός ο χρόνος θα πρέπει να διατηρηθεί στενός, παρόλο ότι αναγνωρίζω και ομολογώ πως θα πρέπει να εξακολουθεί να εφίσταται. Δεν θα πρέπει όμως να φτάσουμε σε ένα σημείο που ε, να είναι διαθέσιμο στους πολίτες μόνο το τελευταίο ε, στάδιο των ε, εγγράφων. αυτό δεν θα βοηθάει τους πολίτες να συμμετάσχουν στη λήψη των αποφάσεων. Μετά, προστασία των δεδομένων και διαφάνεια. Υπογραμμίζω την συνένεση ο Ευρωπαίος τη συνένεση του, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και του ε, Επιτρόπου προστασία, του, ε, Ελεγκτή Προστασίας Δεδομένων. Ε, επίσης υπογραμμίζω ότι η Σύμβαση Άρχους για την προστασία των δεδομένων περιβαλλοντικής φύσεως απαιτεί αλλαγές στον κανονισμό τα όργανα δεν έχουν συμμορφωθεί με την σύμβαση του ο Άρχους. Επίσης αναφέρω ότι οι διεθνείς σχέσεις δημιουργούν καινούριε προκλήσεις, καινούρια προβλήματα και λέω ότι έχει έρθει η στιγμή να ε, ανοίξει, να γίνει πιο προσβάσιμη η λήψη αποφάσεων για θέματα διεθνών διαπραγματεύσεων. Ε, ως ε, θεσμικό όργανο έχουμε ε, επικρίνει στο παρελθόν το Συμβούλιο και, τον, και την ε, Κομισιόν ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, για παράδειγμα, σε διαπραγματευτικές εντολές για διεθνείς συμφωνίες. Επίσης αναφέρω την αρχή της καλής διακυβέρνησης που απαιτεί να διαθέτουμε ένα ενίο δίκαιο για την ε, διοικητική δράση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, ελήψη τέτοιου είδους κανονισμού δεν, τυχάνουν δεν εγγύηση στα δικαιώματα των πολιτών για πρόσβαση στα έγγραφα και τις πληροφορίες. Αυτά. Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα ανοίξει λίγο περισσότερο τις συζητήσεις μας και για την έκθεση Κάσμαν, γιατί εξετάζοντας το πόσο εφαρμόζεται ο κανονισμός, ποια είναι τα προβλήματα τα στην εφαρμογή του, ποιες είναι οι απαιτήσει για αλλαγές, τροποποίησεις των, ε, στους κανονισμούς, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να φτάσουμε σε ένα συμβασμό. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αναβάλουμε άλλο την, ε, ε, τη σύνταξη του κανονισμού. Έχουμε ήδη καθυστερήσει και βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ας δούμε τι έχουν να πούν τα μέλη. κυρία Σόμνερ έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όντως είναι στενά συνδεδεμένη με την έκθεση Κάσμαν η έκθεση κυρίας Χάουτ. Είναι μια καλή έκθεση μια καλή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε ασφαλώ. Κάποια σημεία τα θεωρούμε ευπρόσδεκτα, κάποια άλλα για μένα είναι ακόμα κάπω ασαφή και χρειάζονται περισσότερε διευκρινήσει. Φέρει Στην, ε, στο αιτιολογικό σημείο Γ και μετά επανέρχεται στο 20 αναφέρεται το κείμενο στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, στη διαδικασία λήψη αποφάσεων ω δυνατό περιορισμό της διαφάνειας. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ρητή αναφορά με συνθήκες. Επίσης, σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκε στι αιτιολογικέ ε, προτάσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι ε, εν γέννη έγγραφα ευαίσθητα, έγγραφα δηλαδή τα οποία δεν είναι διαθέσιμα ε, πάντοτε στο ευρύ κοινό και γι' αυτό δεν μπορούμε να στήσουμε να ισχύουν οι κανόνες διαφάνειας. Στο σημείο 41 επίσης ε, δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ. Υπάρχουν προτάσεις. Στο ένα επανέρχομαι με το αίτημα για γενικές αρχές ταξινόμησης ή όρους ταξινόμησης με, τη μορφή κανονισμού ε, που ήδη, οι κανόνες διαβάθμισης ήδη πιστεύω ότι έχουν καλυφθεί από μια σχετική συμφωνία, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Επίσης ε, η παραπομπή στο σημείο 12 σε μια σε μια πρόταση για ένα φιλόδοξο νέο νόμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελευθερία τη πληροφορία. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη στην έκθεση Κάσμαν. σω πάλι να χρειάζεται επαλήθευση. Και επίση γιατί. Ε, θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιο γιατί είναι η πρόσβαση στα έγγραφα θεμελιώδε δικαίωμα. Εγώ βέβαια πάντα είμαι υπέρ της ε, ελεύθερης προς τα δικαιώματα αλλά, στα έγγραφα, αλλά το να ταξινομούμε αυτή την ιδέα, αυτή την αρχή στην κατηγορία των θεμελιωδών ελευθεριών είναι νομίζω περιβολικό. Επίσης από την έκθεση βρίσκω θετικό το ότι υπάρχει μια πρόταση για space to think. Είναι κάτι το οποίο νομίζω έχουμε πακίως επαναλάβει και υποστηρίξει στις συζητήσεις μας. Δεν μπορούμε βέβαια πάντα να ε, επιτρέπουμε την πρόσβαση του κοινού σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων και σε κάθε θέμα, διότι εάν είναι έτσι ε, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε στα τη δουλειά μας, θα είμαστε δηλαδή ε, δέσμοι και δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Πιστεύω όμως ότι αυτές τις επιφυλάξεις η κυρία Χάουτολα θα τις λάβει υπόψη. Για τη τελευταία ανάλυση ξεχνάμε ότι κάθε είδους συζήτηση την οποία πραγματοποιούμε εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο οδηγεί σε μια λήψη απόφαση. Άρα θα μπορούσε κάθε είδου συζήτηση να χαρακτηριστεί ω βάση λήψη αποφάσεων ή διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και γι' αυτό καλό θα ήταν να μην ε, αφήσουμε πεδίο ανοιχτό, ούτε βέβαια για ε, χωρίς κανένα περιορισμό πρόσβαση, αλλά ούτε και για ενδεχομένως απόλυτο αποκλεισμό του κοινού από κάθε είδους έγγραφο. Παρακαλώ λοιπόν με περισσότερη προσοχή να σταθμίσουμε τα πράγματα. Ε, κατά τα άλλα, βέβαια, σαν αρχή η πρόσβαση στα έγγραφα και εγώ 12 χρόνια που είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω συνηθίσει στην ιδέα του να είναι ε, τα έγγραφά μα δημόσια κτλ. Και, και δεν μπορούμε βέβαια να δεχθούμε την υπόνοια ότι ενδεχομένω όλοι οι βουλευτέ ή κάποιοι είναι τρομοκράτε και γι' αυτό πρέπει να ε, χαρακτηρίζονται ω απόρριτα τα σχετικά έγγραφα. Είμαι λοιπόν γενικά υπέρ τη αρχή και η διαφάνεια που ισχύει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ισχύει και στα λοιπά όργανα. Ε, έγγραφα από τον τριμερή διάλογο και από τι διαδικασίε συνδιαλλαγή επίση. Λέτε να είναι και αυτά προσβάσιμα στο κοινό. Προσοχή! Διότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποτυχία πολλών από τι διαδικασίε διαπραγματεύσεων και συνδιαλλαγή που έχουμε. Και δεν ξέρω καν αν θα είναι δυνατόν να γενικεύσουμε τον κανόνα έτσι ώστε να ισχύει σε κάθε τριμερή διάλογο, γιατί ο κάθε ένας από τους τριμερείς διαλόγους ανάλογα με το θέμα έχει διαφορετική έκβαση. Και επισημαίνω επίσης ότι εάν ε, ισχύσει αυτός ο κανόνας της ε, δημοσιοποίησης κάθε είδους εγγράφου που εμπλέκεται στον, ε, στη διαδικασία της διαλλαγής του τριμερή διάλογο, δεν θα μπορούμε να απαλλαγούμε από τις πιέσεις των λόμπι. Θα είναι διαρκώς μπροστά μας. Συνεχίζουμε το σημείο 32 και το αίτημα για ε, κυρώσει σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους κύρωση, συνέπεια, αλλά πρακτικά πώς θα εφαρμοστεί αυτό δεν είμαι βεβαία. Στο D32 θέσπιση νέων θέσεων ειδικά εκπαιδευμένων υπαλλήλων ε, ώστε να δημιουργηθεί βέλτιστη δυνατή προορατική πολιτική Δεν πρέπει να λησμονούμε εδώ όμω ότι η κάθε υπηρεσία, το κάθε όργανο έχει το δικαίωμα να επιλέγει το δικό του προσωπικό και να προσδιορίζει την, ε, τις δραστηριότητες του και το πεδίο δραστηριοτήτων που θέλει. Στη συνέχεια, εκεί όπου γίνεται πάλι λόγος για τις εργασίες των εσωτερικών οργάνων του Κοινοβουλίου και των βουλευτών, θα ήμουν επίσης πολύ επιφυλακτική. και όπως είπα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου πρέπει να, είμαστε, να εργαζόμαστε σε συνθήκες απορρίπτου ή εμπιστευτικότητας για να μπορούμε να κάνουμε πραγματικά καλά τη δουλειά μας. Επίσης ε, προς το τέλος ε, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα πρέπει η πρόσβαση στα έγγραφα για το κοινό να μην αναμειγνύεται με αυτήν της ε, διοργανικής πρόσβασης στα έγγραφα που πιστεύω έχουμε επιλύσει με την έκθεση Cashman. Και χωρίς να θέλω να είμαι υπεραισιόδοξη, Πιστεύω ότι με τι παρατηρήσει αυτέ που έκανε, εφόσον ληφθούν υπόψη, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε με τη συνάδελφο κυρία Χάουταλα σε, μια καλή, ε, σε ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαι βεβαία ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία και απλώ έχουμε μερικά πράγματα ακόμη να διευκρινίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. Ένα σχόλιο να κάνω. Σχολιάσατε την επάρκεια όσον αφορά το θεμελιώδη δικαίωμα όσο τα έγγραφα. Θα ξέρετε ότι η θεωρητική κατηγορία των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν έχει παγιωθεί σε κάθε νομικό σύστημα των διαφόρων κρατών μελών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον είναι γεγονός ότι αυτή η κατηγορία θεμελιωδών δικαιωμάτων όπου υπάρχει, υπάρχει διαφορετική έχει διάφορες προδιαγραφέ στα διάφορα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Έχουμε Ευρωπαϊκή Χάρτα όμως θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχει θεσπίσει επακριβώς το δικαίωμα της προσβάσεως στα έγγραφα. Στο άθρο 42 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλεί τον καθορισμό τον ορισμό ενός συγκεκριμένου θεμελιωδούς δικαιώματος σε κάποιο νόμο σύστημα, όπως το συνταγματικό δίκαιο της Γερμανίας, της Ισπανίας. Λέει ότι είναι δικαίωμα γενικό, το οποίο αναγνωρίζεται, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και απορρέει το γεγονός ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Ότι είναι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσης και συνεπώς είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες τώρα έχουν δικαίωμα στο θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, διότι η Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι ένας από τους πυλώνες από τα συστατικά στοιχεία της συνθήκης της Λισαβόνας. Οπότε είναι εφαρμοστέο δίκαιο. Είναι νόμος. Και γι' αυτό το συζητούμε. βάσει της εκθέσεως της κυρίας Χαουτάλα. Να δούμε τι, έχω, έχει να πει ο συνάδελφός μας, ο κ. Μωράης, που θέλει να πάρει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Μάικλ Κάσμαν απουσιάζει σήμερα, δεν μπορεί να παρίσταται, τον αντιπροσωπεύω εγώ, τον εκπροσωπώ εγώ. Άκουσα τα τελευταία σας σχόλια και αυτά που είπε και η κυρία Σόμερ. Δηλαδή, η ανελευθερία της ενημέρωσης είναι θεμελιώδης δικαίωμα εγώ πώς τα εκλαμβάνω. Πώς εκλαμβάνω την προσέγγιση του κ. Κάσμαν για τον κανονισμό 1049, ότι πρέπει να υποθέσουμε ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία ενημέρωσης και προσβάσεως στα έγγραφα και μετά θα συζητήσουμε τις εξαιρέσεις. Αυτή ήταν η προσέγγιση του. Και αυτή θα είναι η προσέγγιση που θα ακολουθήσει και η έκθεση της κυρίας Χάουταλα. Οι τροπολογίες που θα υποβάλει, θα υποβάλει του Μάικλ και σαν ομάδα θα αφορά τις εξαιρέσεις από τον κανόνα. Και ο κανόνα θα είναι η ελευθερία της ενημέρωσης, ε, που έχει πρωταρχική σημασία. Ο Μάικλ ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα την Χάιντι Χάουταλα για την πολύ ενδελεχή ε, έκθεσή της, υποστηρίζει πλήρως την προσέγγιση της και θα εξετάσει πόσες συστάσεις μπορεί να συμπεριλάβει στην αναθεώρησή του για τον κανονισμό 1049. Σαν ομάδα καλωσορίζουμε την ε, αναφορά του συνταγματικού πλαισίου ε, της θεσμικής διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ενώσης που αναφέρει θήκη της Αβώνας και τις παραπομπές σε συγκεκριμένη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπως την περίπτωση της ε, βαβαρικής μπύρας και την πρόσφατη υπόθεση Info Europe θεωρεί ο κ. Κάσμαν και πιστεύει ότι αγνοήθηκαν αυτά στην πρώτη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 και στη δεύτερη της ε, πρόταση του Μαρτίου του 2011. Αν ήταν εδώ θα ζητούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει εκ νέου γιατί έχει δύο συνυπάρχουσες προτάσεις που αφορούν τον ίδιο κανονισμό. Συμφωνεί η ομάδα μας ότι οι κοινοί κανόνες ταξινομήσεως των εγγράφων, διαβαθμίσεως των εγγράφων και ο καθορισμός του εγγράφου πρέπει να αποτελεί, είναι θέμα που αποτελεί προτεραιότητα, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλα όργανα και θα πρέπει να διευκρινιστεί στην νομοθετική αναθεώρηση. Τέλος, όσον αφορά την προσέγγιση του κυρίου Κάσμαν, θα εξετάσει προσεκτικά το έργο της κυρίας Χάουταλα να δει τι συστάσεις μπορεί να συμπεριλάβει, να λάβει υπόψη και την ευχαριστή εκ νέου για το έργο της. Σας ευχαριστώ κύριε Μόραες. Υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο, άλλος βουλευτής που επιθυμεί να σχολιάσει. Ας επιστρέψουμε στην κυρία Χάουταλα να συνοψίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αισθάνομαι πολύ αισιόδοξη. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και να λύσουμε και τα εκρεμή ζητήματα της εκθέσεως Κάσμαν και πιστεύω ότι ο κύριος Κάσμαν εκ μέρους όλων των σκιωδών εισηγητών μας ζήτησε μια συνεδρίαση με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς που είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ώστε να επιτευχθεί συμφωνία περί υποστηρίξεω από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής των προσπαθειών του Κοινοβουλίου στο συγκεκριμένο ζήτημα που καλύπτεται από την έκθεση του κυρίου Κάσμαν ε, και τη δική μου προσέγγιση. Πράγματι μπορούμε σιγά σιγά να μειώσουμε τις εσωτερικές μας διαφορές και να δούμε κάποια συγκεκριμένα σημεία που εκκρεμούν. Δύο βασικά ζητήματα τίθενται νομίζω. Πρέπει να επεξεργαστούμε αυτό, αυτή την έννοια του χώρου ανάλυσης, σκέψης αν θέλετε. Ε, όλες οι ανταλλαγές, οι γραπτές πρέπει να είναι δημόσιες. Ε, χρειάζεται κάποια διαχωριστική γραμμή μεταξύ υπομνήματος ανεπίσημου εγγράφου και πότε αυτό γίνεται επίσημο δημόσιο έγγραφο. Αυτό μπορεί να καθοριστεί. Μετά ε, πρέπει να δούμε του πώς θα πρέπει να εφαρμόσουν διάφορες, διάφοροι κανόνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα μέλη αυτού. Ε, πιστεύω ότι έχουμε σωστό νόμο που προστατεύει την ιδιωτική ζωή και μπορούμε ίσως να εργαστούμε βάσει της εξής υποθέσεως για τους ευρω... αποζημιώσεις και δαπάνες των βουλευτών όσον αφορά την χρήση χρημάτων του φορολογωμένου, το θέμα τη δικαιώματο του κοινού να έχει πρόσβαση στα έγγραφα. Πρέπει να εφαρμόζεται αυτό. Αλλά δεν θεώρησα ποτέ ότι κάθε μέλος χωριστά θα πρέπει να παρουσιάζει τις εσωτερικές του, του, εσωτερική του αλληλογραφία, email κλπ. Αυτό αποκλείεται. Πρέπει να βρούμε διαχωριστική γραμμή όσον αφορά το δικαίωμα του κοινού να γνωρίζει για τις δραστηριότητε μας και τις δαπάνες μας. Και πώς αυτό συσχετίζεται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής που έχουμε και εμείς αυτό το δικαίωμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά άλλα εκρεμή θέματα και προσβλέπω στις συνομιλίες μου με τους κοιόδης ηγητές όποτε αυτό θα είναι δυνατόν, το συντομότερο δυνατόν. Καλώς, πριν πάμε στο επόμενο σημείο, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Συμβούλιο θέλουν να πούν κάτι. Έχουμε παρόντες εκπροσώπους τους. Θέλετε να πείτε κάτι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορίστε, έχετε το λόγο. Sorry. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να διατυπώσω πολλά σχόλια αυτή τη στιγμή. Απλώς πολλές από τις συστάσεις της εκθέσεως θα επισημάνω ήδη εφαρμόζονται. αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα η πρόσβαση στα δικαιώματα, στα έγγραφα και όχι μόνο τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και νωρίτερα από το Άμστερνταμ ήδη είχε εδρεωθεί και δεν υπάρχει αμφιβολία προς το ότι είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Για την εφαρμογή του κανονισμού δεν αμφισβητείται ποτέ ότι δίποτε αιτήματα σε πρόσβαση μάλλον ε, σε αποκλεισμό από την πρόσβαση θα πρέπει να στηρίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες εξαιρέσεων. Αυτό ισχύει πάντα για την Επιτροπή. Μόνο βάσει εξαιρέσεων επί του κανονισμού μπορεί να αποκλείσουμε την πρόσβαση στα δικαιώματα. Μπορεί αυτό βέβαια να οδηγήσει συζήτηση προς το πεδίο ε, και την εφαρμογή του πεδίου του κανονισμού, αλλά εμείς όπως είπα μόνο εξαιρέσεις που ισχύουν για τον κανονισμό ρητά εφαρμόζουμε για την για τον περιορισμό της πρόσβασης. Το space to think σημαίνει όχι μόνο νομοθετική διαδικασία, αλλά και γνωστή ε, ε, και την μη νομοθετική διαδικασία. Αυτή δηλαδή τη διαδικασία, το space to think, τη χρησιμοποιεί η Επιτροπή κυρίω όχι για την νομοθετική διαδικασία, αλλά για τη μη νομοθετική, δηλαδή τι διοικητικέ διαδικασίε, την ε, προεπεξεργασία. Επίση, λαμβάνεται πάντα υπόψη ε, το γεγονό ότι σχετίζεται με την ε, ευρύτητα της Δημοσιοποίηση των εγγράφων, δηλαδή μέχρι ποιο βαθμό έγγραφα μπορούμε να φτάσουμε. Θα φτάσουμε μέχρι και τα άτυπα έγγραφα, θα δημοσιεύουμε ακόμη και τα email. εκεί λοιπόν τα πράγματα ε, δυσκολεύουν και πρέπει να εισαγάγουμε ενδεχομένω κάποιους ε, περιορισμούς. Το θέμα λοιπόν το Space Thing έχει εισαχθεί ήδη προς συζήτηση και ακόμη δεν έχει επιληθεί με βάση τον κανονισμό 1049. Αλλά θα ήθελα να εξηγήσω τα εξή. Η πρώτη πρόταση κατατέθηκε το 2008 στι 30 Απριλίου σε μια χρονική στιγμή όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να λάβει υπόψη την υφιστάμενη με αυτό την ομολογία. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο κατηγορεί την Επιτροπή ότι δεν λαμβάνει επαρκώ υπόψη την ομολογία, αλλά η απόφαση Τούρκο, η οποία αναφέρεται συχνά ε, στις ε, αιτιολογίες του εγγράφου, ε, ήταν μεταγενέστερη της πρότασης. Και η Επιτροπή, όπω σα είπα, λαμβάνει υπόψη πάντα όλη την ομολογία και αυτό σημαίνει όλη την ομολογία και όχι μόνο κάποιε συγκεκριμένε ή επιλεκτικέ αποφάσει ε, του ε, δικαστηρίου. Αυτή λοιπόν είναι ακόμα έτσι στην πρώτη ανάγνωση. Εν τω μεταξύ όμως και μετά ε, την θέση εφαρμογή της Συνθήκης Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι δεν μπορούμε να παραμένουμε σε ασυμβατότητα ως προς την εφαρμογή της συνθήκης και άρα προκειμένου να προσαρμοστούμε στους όρους της συνθήκης, άρθρο 15 παράγραφος 3, ε, προτείνουμε την αυτή, ε, το νέο αυτό σχέδιο κανονισμού. Το 1049 ούτως ή άλλως καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό οργάνων, αλλά δεν καλύπτονται και όλα τα, δεν καλύπτονται 100% όλα τα όργανα και οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή αποκεντρωμένε υπηρεσίε κτλ. Το 1049 έχει μάλλον οριζόντια εφαρμογή. Και επίση υπάρχουν κάποια κενά φερρυπίν ω προ την πρόσβαση στα, για το κοινό στα έγγραφα του ελεγκτικού συνεδρίου που έχει αποκλειστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεωρήσει ότι θα έπρεπε αυτή η νέα και περιορισμένη έκταση πρόταση να κατατεθεί προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν μέγιστη ευθυγράμμιση με τους όρους της συνθήκης. Ο Όμπουτσμαν μάλιστα το είχε προτείνει, έγινε μια συζήτηση με την υπηρεσία του και την Επιτροπή πέρυσι και ο Όμπουτσμαν μας σχεστεί σε αυτές τις ελάχιστες ακόμη αλλαγές. Δεν έχουμε ακόμη αποσύρει την προηγούμενη ε, πρόταση, παραμένει δηλαδή το πεδίο για διαπραγμάτευση με βάση την παλαιότερη πρόταση, αλλά πάντως τώρα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να ευθυγραμμιστούμε στους όρους συνθήκες όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Το Συμβούλιο παρακαλώ. Θέλει να κάνει σχόλια. Καλώς. Θα περάσουμε τότε στο επόμενο θέμα. Ε, σας ενημερώνω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 30 Μαΐου, 30 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα πάω στο επόμενο θέμα που είναι μια συλλογική προσέγγιση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κύριος Μωράης. Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μία σύντομη παρέμβαση για να επισημάνω ότι δεν υπάρχει διερμηνία ε, στα Σουηδικά και η συνάδελφος η οποία έχει αναλάβει τη σκιώδη εισήγηση θα μπορέσει να μιλήσει τη μητρική της γλώσσα διότι δεν υπάρχει διερμηνία από υπρός. Ξέρω ότι έχουμε περιορισμού στην αίθουσα αυτή, έχει συμβεί πολλές φορές, να μην προσφέρεται η, η σουηδική διερμηνία, αλλά παρακαλώ όταν έχουμε συναδέλφους που έχουν λάβει ως χειώδεις συγητές ή ως συγητές ακόμη εκθέσεις, να μεριμνείτε έτσι ώστε να προβλέπετε η γλώσσα τους. Παρακαλώ αυτό να λαμβάνετε υπόψη. Ορθώς λέει ο Πρόεδρος, έχετε πολύ το δίκιο κύριε Μωρές. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία με τον τρόπο αυτό να ε, γύρω και εγώ αυτές τις παρατηρήσεις ως πρόεδρος. Η μόνη αίθουσα που είχαμε στη θέση μας για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν ακριβώς η αίθουσα όπου βρισκόμαστε τώρα με τις 12 καμπίνες, 12, ούτε μία παραπάνω, και επίσης ε, πρέπει να επισημάνω ότι έγινε μια επιπλέον προσπάθεια για τα ουγγρικά στο 6, τα ρουμανικά στο 10, τα πολωνικά στο 11 και τα σλοβενικά στο 12. Έτσι, ναι, μεν, έχετε δίκιο ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα για όλες τις γλώσσες, λόγω ακριβώς της ε, διευθέτησης των ε, χώρων σε αυτή την αίθουσα. Βεβαίως και έχουν δικαίωμα οι βουλευτές να χρησιμοποιούν ε, και να ακούν τη γλώσσα τους, μια επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για λόγους επιμελητιακούς δεν είναι πάντοτε δυνατόν να προσφερθούν σχετικές υπηρεσίες, όπως συμβαίνει και τώρα. Και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Σας βεβαιώ ότι αυτό συμβαίνει μόνο σε όλες έκτακτες περιστάσεις και όταν έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα, τέτοια προβλήματα. Η κυρία Ζόμερ. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, μια σύντομη παρέμβαση. Δεν είναι όλος εξαιρετικέ περιστάσεις στις οποίες ε, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι, σήμερα βλέπουμε ότι είναι γεμάτες όλες οι καμπίνες. Πολύ καλά. Αλλά εγώ διαπιστώνω ότι στην Επιτροπή μας δεν έχω τη δυνατότητα πάντοτε να έχω τη μητρική μου γλώσσα. Δεν υπάρχουν πάντοτε τα, γράμματα, τα έγγραφα. Πολλές φορές στις τροπολογίες ακόμη, οι αντίστοιχες ε, προτάσεις δεν τις βλέπω στη μητρική μου γλώσσα και είμαι υποχρεωμένη να λαμβάνω αποφάσεις χωρίς να μπορώ να διαβάσω το κείμενο όπως ε, θέλω στη μητρική μου γλώσσα. Και αυτό δεν ξέρω αν σημαίνει ότι δεν γίνονται επαρκοκέεις προσπάθειες ή εάν τελικά ε, είμαστε τόσο πολύ... Έχουμε τόση πολλή δουλειά που η γραμματεία δεν προλαβαίνει να βγάλει την δουλειά που χρειάζεται. Και ρωτώ, Πρόεδρε, γιατί δεν παρεμποδίζετε εσείς, σε επίπεδο Επιτροπής, την παραγωγή ε, ε, τέτοιου όγκου δουλειάς που μας οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δουλεύουμε σε αυτήν την επιτροπή όπως μπορούμε, όπως θα θέλαμε καλύτερα, διότι δεν έχουμε σχεδόν ποτέ, ποτέ τη μετάφραση στις τροπολογίες μας, στις εκθέσεις μας. Εδώ με την έκθεση της κυρίας Χάουτα Αλαφερυπίν. 30 Μαΐου έχετε ορίσει την προθεσμία, 15 τι ψηφοφορίε. Φυσικά και θα προλάβει η μετάφραση να έχει τι τροπολογίε έτοιμες σε όλες τι γλώσσες. Άρα και εδώ πρόκειται για μια βασική ε, τοποθέτηση που πιστεύω θα πρέπει να ρυθμιστεί. Και οι συνάδελφοι συντομιστέ ε, και το Προεδρείο της ομάδας ε, αλλά ασφαλώ και ο κάθε βουλευτή όπω εγώ ίδια δεν μπορούμε να δουλεύουμε σωστά όταν δεν έχουμε τα έγγραφα στη θέση μα. Ασφαλώ. Έχετε δικαίωμα ελέγξω λίγο την κατάσταση ε, ζητώντας από τους ε, συντονιστές και από τους εισηγητές να κάνουν τη δουλειά τους έτσι ώστε να βοηθήσουν ε, όλη την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με ένα ορθολογικό τρόπο την ημέρηση διαταξή της. Παρόλες τις προειδοποιήσεις, πολιτικές ομάδες και μέλη εξακολουθούν να πιέζουν όχι μόνο για νομοθετικά θέματα αλλά και για ε, ιδέες πρωτοβουλίας νομοδοτήσεις. Ε, υποβάλλουν ιδέες, ε, πολυάριθμες ιδέες οι οποίες δημιουργούν βέβαια και ένα μεγάλο όγκο εγγράφων τα οποία θα πρέπει να μετα φράζονται κλπ. Κάτι που δημιουργεί πραγματικά σημαντικό πρόβλημα στις υπόλοιπες ε, υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως στις συναντήσεις συντονιστών ε, έχω επιστήσει την προσοχή σε όλα τα μέλη, ε, την προσοχή τους ε, για αυτό το ε, καθόδες θέμα. Δυστυχώς όμως εγώ ως πρόεδρος δεν μπορώ από μόνος μου να αποθαρρύνω τα μέλη ή τις πολιτικές ομάδες από το να υποβάλουν αυτές τις ιδέες. Νομίζω ότι η κατάσταση αυτή μας αφορά όλους. Το σημειώνω, αλλά ε, σίγουρα το σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα ε, και όσο πιο πολύ το συνειδητοποιούμε τόσο πιο πολύ θα λύνεται το πρόβλημα. Πρέπει να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας με υπευθυνότητα. Θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο ή θα συμφωνήσετε με την κυρία Σάμερ. Ε, κύριε Σκίφλερ, είμαι πρόεδρος τη Επιτροπής Ανάπτυξης, έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Ε, το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση με τους προέδρους και τους συντονιστές για να βρούμε μια λύση. Γιατί στην επόμενη θητεία το πρόβλημα δεν θα εξαφανιστεί από μόνο του. Συνεπώς θα πρέπει μια για πάντα να βρούμε μια μόνιμη λύση. Το σημειώνω και αν θέλετε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, εντάξει. Σημείο 5. Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον συνάδελφο Άξελ Βος ως Έχει ήδη γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες που που ε, υποβλήθηκαν στο προσχέδιο της ε, έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας. Ο κύριος Φως θα πάρει το λόγο και μετά έχουμε χρόνο για συζήτηση. Σας ανακοινώνω πάντως ότι η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή θα λάβει χώρα στην ε, συνάντησή μας του Ιουνίου, 15 και 16 Ιουνίου συγκεκριμένα. Και Φως, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε για την αναβολή ε, στις 15 και 16 Ιουνίου της ψηφοφορίας και έτσι έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες. Υπάρχουν δύο λόγια αυτήν την αναβολή. Καταρχά η Επιτροπή ε, μα ευνηδίασε τον Απρίλιο ορίζοντα ένα χρονοδιάγραμμα για το νομοθέτημα αυτό κάπου στα μέσα Ιουλίου, πιο νωρί από, ό,τι από ό,τι είχαμε προβλέψει, ως εκ δεν ήταν δυνατόν να τηρήσουμε τι προθεσμίες και προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε μέσα στο Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουμε το έργο μα από πλευρά μα και να λάβουμε τις σχετικέ ε, ψηφοφορίε, αλλά δεν μπορέσαμε ε, να είμαστε έτοιμοι και έτσι με την αναβολή αυτή μπορούμε να έχουμε πιο πολύ άνεση χρόνου. Βέβαια, ε, οι συνάδελφοι από τις ε, συναρμόδιες για γνωμοδότηση επιτροπές δυστυχώς πιέστηκαν ίσως περιτά. Δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε προκαταβολικά ότι θα αναβληθεί, όπως είπα, η ψηφοφορία. Δεν ήταν γνωστά όλα αυτά και δεν ήταν ορατά από το WebScan. Πάντως ευχαριστώ τους πάντες για τη συνεργασία τους στην υπόθεση αυτή. 155 ήταν οι τροπολογίες που έχω κατατεθεί για την έκθεσή μου. Έχουμε και τις τέσσερις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού Νομικών Ιστορικής Αγοράς και Βιομηχανίας που θα πρέπει επίσης να ενσωματώσω στο κείμενο και εν τέλει διατυπώνοντας και την ε, ικανοποίησή μου για το γεγονό ότι τόσοι πολλοί συνάδελφοι συνέπραξαν στην υπόθεση αυτή, θα ήθελα να ενημερώσω ότι σκοπεύω να καταθέσω συμβαστικές τροπολογίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Είχα και εγώ κάποιες παρατηρήσεις ε, που θα ήθελα να καταθέσω με τροπολογίες ε, και που λόγω περιορισμού χώρου δεν μπόρεσα να ενσωματώσω στο, στο, στο σώμα της έκθεσης. Και θα ήθελα να αναφέρω συνοπτικά ε, την ε, ουδετερότητα ως προς την τεχνολογία, την ε, ελευθερία της γνώμης, την ελευθεροτυπία, την οδηγία για την προσωπική η ζωή, την προστασία του ιδιωτικού βίου, για τις αρμοδιότητες της ομάδας εργασίας 29 και άλλες σημαντικές πτυχές που περιέχονται σε πολλές από τις τροπολογίες είναι επίσης η προστασία των ευάλωτων προσώπων, των μη προστατευομένων, ιδιαίτερα των παιδιών ή των ηλικιωμένων. Είχαμε επίσης πολλές τροπολογίες σχετικές με το θέμα της ασφάλειας και της ελευθερίας, στάθμιση δηλαδή μεταξύ προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων και καταπολέμησης τρομοκρατίας. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην ε, ε, διατύπωση, γιατί ε, τόσο η ασφάλεια όσο και η προσωπική ζωή είναι θεμελιώδη δικαιώματα και θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να διατυπώσουμε το σχετικό κείμενο έτσι ώστε να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ του ε, θεμητού αλλά και του νομικά εφικτού. Βεβαίως το δικαίωμα στην προστασία του ιδιωτικού βίου είναι ανώτερο των άλλων δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει να βρούμε, πιστεύω, μία στάθμη τέτοια που να μην υποχρεώνει κανένα να επιλέξει μεταξύ ασφάλειας και προσωπικής ζωής, ώστε να είναι υλοποιήσιμα δηλαδή και τα δύο αυτά αγαθά ταυτόχρονα. Σκοπεύω επίσης ε, τις επόμενες εβδομάδες να ξανασυναντήσω τους σκιώδεις ηγητές για να συζητήσουμε, για να διευκρινίσουμε ορισμένα σημεία που πιστεύω θα ε, ε θα μπορέσουμε στη συνέχεια να ενημερώσουμε και οδησηγητές τι ομάδε τους ε, για τα σημεία αυτά και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε ε, στη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν μήπως κάποιοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κ. Λαμπρινίδης πρώτος. Είναι πολλές οι τροπολογίες όπως είπε ο Άξελ θα πω τα εξή εν συντομία. Έξοχη είναι η έκθεση του Άξελ. Βασίζεται επί εξόχου προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δουλειά μας είναι να καταλήξουμε σε κάτι καλό. Αυτές πρέπει να πω ότι είναι πολλές τροπολογίες και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον Άξελ και όλους τους κοιόδης εισηγήτες για τις συναντήσεις που είχαμε και για την έξοχη συνεργασία και το συντονισμό. Θέλω να ενθαρρύνω, παρόλο που καθένας έχει δικαίωμα να υποβάλει τροπολογίες, θέλω να ενθαρρύνω παρόλα αυτά τα μέλη να προσπαθήσουν εν γέννη, όχι μόνο αυτή την εκθέση, να έρχονται σε επαφή με τους κοιόδεις των ομάδων πριν υποβάλουν τροπολογίες για να αποφευθεί πολλή δουλειά και να μην υπάρχει επικάλυψη. Βλέπω πολλές τροπολογίες που ήδη καλύπτονται από τροπολογίες των σκιωδών ή θα μπορούσαν να συζητηθούν περισσότερο και να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά το πλαίσιο των τροπολογιών, συμφωνώ με τον Άξελ. Διάφορα ζητήματα σημαντικότατα για μας. Το βασικό θέμα του κανονισμού ή της οδηγίας δεν έχει επιληθεί. Πολλοί θέλουμε οποιαδήποτε λύση βρεθεί να είναι σε υψηλό επίπεδο προστασίας. Το ίδιο ισχύει και για την αυτορύθμιση του τομέα. Καλό αυτό, αλλά σαν συμπληρωματικό μέτρο κατά την άποψή μου όσον αφορά του, της νομοθεσίας. Η αυτορύθμιση αυτή καθεαυτή στον τομέα αυτό που είναι πολύ ευαίσθητος δεν αρκεί. Δεν αποκλείεται βέβαια. Σαν συμπλήρωμα όμως της νομοθεσίας και της νομοθεσίας που εδράζεται επί υψηλών προδιαγραφών. Πέραν αυτού θα συνεργαστώ με τον Άξελ Βος και τους άλλους κοιώδεις ούτως ώστε στο τέλος να έχουμε την, τον πληρέστερο και ευκολότερο κατάλογο ψηφοφοριών όταν έρθει η στιγμή της ε, ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ιντεφελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σημασία του θέματος αυτού κατέστη σαφής για μία ακόμη φορά τις τελευταίες εβδομάδες. Ή ε, το θέμα της το εντοπισμού της Apple, το PlayStation, το TomTom, όλα αυτά τα συστήματα έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύω τα δεδομένα και πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα στη ζωή μας. Αλλά είναι, ήρθε πολύ έγκαιρα αυτή η πρόταση. Και εγώ όπως ο Σταύρος Λαμπρινίδης ευχαριστώ τον εισηγητή για τη συνεργασία μας για την προσέγγιση που ακολούθησα και είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε καλό συμβιβασμό. Νομίζω ότι η προστασία των δεδομένων είναι ευρύτερη έννοια από την απλή προστασία των στοιχείων. Σχετίζεται με προσωπική ελευθερία, το δικαίωμα μη διάκρισης, ισότιμης αντιμετώπισης, σχετίζεται με την επαφή μεταξύ πολιτών και κυβερνήσεών τους ή επαφής πολιτών δημοσίων αρχών είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από απλή τεχνική προστασία των δεδομένων. Σε πρώτερες συζητήσεις τόνισα τρεις διαστάσεις που θεωρώ ότι είναι οι βασικότερες. Και υπάρχει συμφωνία νομίζω στο Κοινοβούλιο από αυτό αλλά και συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε ενιαίες προδιαγραφές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Να συγχωνεύσουμε τους πρώτερους πρώτων και τρίτο πυλών. Αυτό είναι σημαντικότατο. Δεύτερον, χρειαζόμαστε εναρμόνιση. Αυτό θα είναι προς όφελος όχι μόνο της βιομηχανίας, του τομέα, αλλά και των των αντικειμένων μάλλον της χρήσεως. Χρήστες, πολίτες. Μετά τρίτο θέμα, εφαρμογή του νόμου. Έγιναν πολλές καλές προτάσεις, υπέβαλα και εγώ κάποιες ε, τροπολογίες. Ζητώ αυστηρότατες κυρώσεις. Αν γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να προβλέπονται και σημαντικότατες σοβαρότητες κυρώσεις για εκείνους που ε, κάνουν κατάχρηση αυτών των στοιχείων. Κακή χρήση αυτών. Προσβλέπω λοιπόν στις συμβαστικές προτάσεις που θα υποβάλει ο και είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομος και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον εισηγητή Νομίζω ότι είχαμε πολύ καλή συνεργασία και πρόοδο μέσα από τις συναντήσεις με τους σκιώδεις ηγητές. Πολλές από τις ε, τροπολογίες μπορέσαμε να τις διατυπώσουμε από κοινού και έτσι να βελτιώσουμε συνολικά το κείμενο. Και να διευρύνουμε σε έναν βαθμό και το πεδίο αναφορά του. Πράγμα το οποίο θεωρώ ευπρόσδεκτο. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι η ενιαία διαμόρφωση ε, συνθήκων, προδιαγραφών μάλλον προστασίας των προσωπικών δεδομένων ε, είναι πολύ σημαντική και αντιμετωπίζει πιστεύω το πρόβλημα του κατακαιρματισμού μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών ε, μέσων, νομοθετημάτων δηλαδή, που εισάγουν διαφορετικά επίπεδα και αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έτσι λοιπόν η οδηγία 9546 είναι για μας το σημείο εκκίνησης. Δεν θέλουμε οπισθοδρόμη σε σχέση με τις υψηλές προτεραιότητες προστασίας των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων από πλευρά του Κοινοβουλίου και δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τον ανταγωνισμό ή σε σχέση με την, ε, προστασία με, την ασφάλεια δεν είναι έννοιες αντικρουόμενες, δεν βρίσκονται σε σχέση ανταγωνιστική, αλλά μπορούν να συνδυαστούν. Μπορεί οι ανάγκες ασφάλειας ή ανταγωνιστικότητας να περιορίζουν κάποιες δυνατότητες, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι μπορούν να καταπνίξουν την ε, ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων και άξελ είμαι υποχρεωμένο να διαφωνήσω μαζί σου. Δεν υπάρχει θεμελιώδες δικαίωμα στην ασφάλεια σε κανένα έγγραφο ε, του σε κανένα νομοθέτημα, σε κανένα έγγραφο ή διεθνή συμφωνία. Γι' αυτό λοιπόν, ε, ενώ υπάρχει δικαίωμα στην προσωπική ε, ζωή και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, νομίζω ότι είναι υπέρτατη αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος που έχει το λόγο. Ε, Πρόεδρε, ένα-δυο σχόλια μόνο. Πρώτον, καλωσορίζω την έκθεση του Άξελ Βος Το κατά πόσον θα πρέπει να, είναι, να ε, διαθέτουμε κανονισμό ή οδηγία επαφείται στην Κομισιόν αλλά είναι ενδιαφέρον. Αν επιλέξουμε τον κανονισμό, ο κίνδυνος είναι ε, να αποδυναμωθεί όπως συμβαίνει πολύ συχνά με του κανονισμούς, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο αποτελεσματικός από ότι μια αυστηρή οδηγία. Σίγουρα πάντα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τέτοιου είδου θέματα, ε, ιδιαίτερα όταν προκύπτουν οικονομικά και διοικητικά άχθη. Και επίσης να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την αναλογικότητα. Για παράδειγμα, με τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων. Ε, τι θα σήμαινε αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, καθώς επίσης και για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μετά, εναρμόνιση πρακτικών Ε, είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Ε, να αναφερθώ στην γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Πολιτισμού για αυτό το θέμα. Δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει να καταρτήσουμε, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σε θέματα προστασίας δεδομένων ως κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος στα σχολεία. Νομίζω ότι αυτό θα δημιουργούσε τρομακτικά, τρομακτικό διοικητικό άχθος. Ίσως θα πρέπει να, τους, να τα εκπαιδεύσουμε πιο πολύ για το ποδόσφαιρο και τους ποδοσφαιριστές και μερικές ε, φορές οι ποδοσφαιριστές παραπέμουν και σε θέματα προστασίας δεδομένων. Ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σύστημα αυτό. Επίσης ε, δεν θεωρώ ότι καλύπτεται το, η περίπτωση συλλογικών προσφυγών για αποζημίωση. Ε, θα πρέπει να δούμε, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς τι θέλουμε να εναρμονίσουμε και μέσα αυτή την εναρμόνιση να δούμε τους βασικούς κανόνες, να είναι πολύ πιο σαφείς αυτοί οι βασικοί κανόνες ο κοινό παρανομαστής. Κατά τα άλλα, καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλία. Έχω υποβάλει τροπολογίες, αλλά συνεργάζομαι πολύ στενά με τον κύριο Βό. Ευχαριστώ. Thank you. Now, Mr. Κύριε Ernst. Καταρχά, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή. Ήταν ε, καλή δουλειά, προέκυψε καλή έκθεση. Ευχαριστώ ιδιαίτερω για την πολύ καλή συνεργασία και τη συζήτηση επί της ουσίας των θεμάτων που ήταν πολύ ικανοποιητική και πιστεύω θα πρέπει να συνεχιστεί με αυτό το τέλος τη συζήτηση ώστε να έχουμε μια καλή έκθεση ως τελικό αποτέλεσμα. Στο πρώτο πράγμα που θα ήθελα να αναφερθώ. Πάντα πρέπει να έχουμε ε, υπόψη ότι το ε, δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι θεμελιώδες δικαίωμα και δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Επίσης, το ίδιο θα πρέπει να αξιολογούμε, με τον ίδιο γνώμα θα πρέπει να αξιολογούμε τις ε, προσβολές του δικαιώματος αυτού. Και γι' αυτό ιδιαίτερα θα ήθελα να υπογραμμίσω τις τροπολογίες εκείνες για την αρκετές οι οποίες σημαίνουν την ανάγκη για την ανάληψη αποτελεσματικών μέτρων σε περίπτωση προσβολής αυτού του δικαιώματος, ώστε να είναι αποτελεσματική η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η, ε, η αποτροπή από παραβιάσεις αυτών. Δηλαδή θέλουμε, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, να είναι αποτελεσματική η νομοθεσία που θα εφαρμόζεται. Μια δεύτερη παρατήρηση. Στην προστασία των προσωπικών δεδομένων πάντα τα επανέρχεται η αρχή, η ιδέα της αναλογικότητας της, του μέτρου της, η τελολογική αρχή ε, και ούτω θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε όταν ορίζουμε τέτοιου είδου νομοθεσία ότι θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος πολίτης να γνωρίζει τι συμβαίνει με τα προσωπικά του δεδομένα που αποθηκεύονται, Φερρυπίν. Θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι σε θέση τα δεδομένα τα οποία την χάνουν επεξεργασία, να ζητήσει και να διαγραφούν και να είναι σε θέση περαιτέρω ο ίδιο να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Εάν τα αφήσουμε αυτά όλα ασαφή, νομίζω ότι η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο εγώ προσωπικώ αποδίδω ιδιαίτερη σημασία. Τελευταίο, ε, τρίτο σημείο, το ζήτημα του ε, διαμεσολαβητή και το επίπεδο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Πιστεύω εδώ ότι έχουμε μπει στο σωστό δρόμο και θα πρέπει, όπως αναφέρετε και εσείς, να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του διαμεσολαβητή για τα προσωπικά δεδομένα. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε στο μέχρι στο δυνατό βαθμό τους πολίτες ε, σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τους νέους και τους ηλικιωμένους, πώς δηλαδή θα πρέπει να χειρίζονται τα θέματα των προσωπικών τους δεδομένων, ε, πώς θα πρέπει να επαγρυπνούν ώστε να μην πέφτουν θύματα παραβιάσεων. Αυτό τόσο για τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους όπως είπα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι έχουμε, ένα, έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ καλό δρόμο. Κύριε Σταβάρης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή μας ε, συνεργάστηκε πάρα πολύ καλά με τους κοιόδης εισηγητές και με τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τα πρώτα βήματα προκειμένου να θεσπίσουμε μια συνολική φιλοσοφία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητη και επίγουσα, διότι μια σειρά προβλημάτων σχετικών με την προστασία των δεδομένων όπως για παράδειγμα η κλοπή ταυτότητας κλπ. ή και άλλα σε σχέση με τα γενικότερα δικαιώματα στην προσωπικότητα, σε ε, μη διάκριση ε, που κάποιοι <clears throat> θεωρούν ότι ε, υπάρχουν όπως και άλλα δικαιώματα που, για τα οποία συζητώνται, τα δικαιώματα στην, το δικαίωμα στην ευτυχία. Ε, για το οποίο κάνει λόγο το Αμερικανικό Δίκαιο. Όλα αυτά έχουν σχέση με την φιλοσοφία προστασίας των δεδομένων την οποία αναζητούμε αυτή τη στιγμή. Ε, η φιλοσοφία είναι βέβαια λίγο αφηρημένη, αλλά η πραγματική ζωή είναι πολύ συγκεκριμένη και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα ε, σε σχέση με το απόρριτο των πληροφοριών μας, ε, τις ε, κλοπές ταυτότητας, της προσβολής της προσωπικής μας ζωής και του προσωπικού μας χώρου. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να καθορίσουμε ε, αυστηρά κριτήρια για την πλαισίωση της προστασίας των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε διαφωνώ με την γνώμη του κ. Κίρκοπ ότι θα έπρεπε να κινηθούμε προς μια οδηγία και όχι προς ένα κανονισμό. Όχι, η οδηγία δίνει πολύ μεγάλο περιθώριο ελιγμών στη μεταγραφή της σε εθνικό επίπεδο, στην εθνική νομοθεσία και επιτρέπει μάλλον αποτρέπει επαρκή εναρμόνιση έτσι ώστε να λάβουμε πρακτικά αποτελέσματα. Πολύ δε περισσότερο που οι μεγάλες βάσεις δεδομένων είναι διεθνείς και διασυνοριακές, ε, το οποίο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια εναρμόνιση, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ένας κανονισμός θα μας επέτρεπε να είμαστε πιο αυστηροί σε ό,τι αφορά αυτήν την εναρμόνιση. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι κύριοι Λαμπρινίδης, Άλμπρεχτ κλπ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το θέμα ε, της ευαισθητοποίησης στα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων. Ε, τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να καθοριστούν με έναν τρόπο σαφή στο πλαίσιο ενδεχομένως μιας χάρτας δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων. Αυτό θα διευκόλυνε τους πολίτες να τα επικαλούνται σε περιπτώσεις που θα παρουσιάζονται διαφορές. Για παράδειγμα, δικαιώματα όπως ε, θα ε, είσαι υποχρεωμένος να, σβήσεις τα προσωπικά μου δεδομένα όταν σου τα ζητήσω. Ε, δεν επιτρέπεται να τα δημοσιοποιήσεις χωρίς την άδειά μου κλπ. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να τα συνοψίσουμε όλα αυτά τα δικαιώματα με έναν τρόπο πολύ σαφή για τους πολίτες, έτσι ώστε να τα γνωρίζουν, προκειμένου να μπορούν να τα προστατεύσουν. Σε, αυτό το πρώτο στάδιο είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο καλή εφαρμογή των αρχών και των ιδανικών που μα εμπνέουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ταβάρε. Αν δεν υπάρχει άλλο που θέλει να μιλήσει... Α, ορίστε, κύριο κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο γιατί εν γέννη συμφωνώ με τον κύριο Βος. Ε, δεν θέλω να σχολιάσω το θέμα του κανονισμού της οδηγίας, αλλά θέλω να κάνω μια μικρή διόρθωση ε, σε ό,τι αφορά την δήλωση του Ζωαν Φιλίπ, ε, στην οποία δεν αντέδρασε κανείς άλλος συνάδελφος. Ακόμα άκουσα ότι είπε, πως είπε ότι η ασφάλεια δεν υπάρχει ως θεμελιώδες δικαίωμα. Θα ήθελα να το διορθώσω και να αντιδράσω αμέσως στο άρθρο 6 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο ακριβώς για αυτό το θέμα. Όλα τα δικαιώματα, όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, λέει. Συνεπώς πρώτα η ελευθερία και μετά η ασφάλεια. Οπότε, Ζωάν Φιλίπ, η ασφάλεια είναι θεμελιώδες δικαίωμα στο άρθρο 6 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχοντας ακούσει αυτή την αναφορά στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Ας δώσουμε το λόγο ξανά στον κύριο Βος, ούτως ώστε να ανακεφαλαιώσει. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρατηρήσεις των συναδέλφων και για να επανέλθω στο τελευταίο αυτό σημείο ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και το ποια είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα ήθελα να επισημάνω ότι στο γερμανικό τουλάχιστον σταγματικό δίκαιο υπάρχει η ιδέα της ε, σύμπραξη, τη συλλειτουργία αυτών των δικαιωμάτων. Συνυπάρχουν δηλαδή, δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Αυτό ισχύει σε διάφορα θέματα. Ε, στις παρατηρήσεις λοιπόν υπήρξαν κάποιες ε, ερωτήσεις, σε ένα βαθμό μάλιστα σε λεπτομέρειες, τις οποίες πιστεύω θα δούμε πιο συγκεκριμένα την ώρα που θα έχουμε την συγκεκριμένη πρόταση και θα πρέπει να συζητήσουμε τι θέση θέλουμε να τηρήσουμε. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα θα πρέπει να ε, επισημάνουμε ότι προσπαθούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα και σε αυτό πιστεύω ότι είναι όλες οι παρατηρήσεις για την προστασία των, απο, των προσωπικών δεδομένων, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το στόχο τίνουμε. Για το θέμα κανονισμός ή οδηγία δεν θέλω να το μετατρέψω σε δογματικό ερώτημα. Ε, το περιεχόμενο με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο και σε αυτό θα ήθελα να επικεντρωθώ. Εάν έχουμε μια σαφή οδηγία, μια οδηγία που είναι διατυπωμένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί του στόχους μας και να φτάνουμε στο επιδεκόμενο αποτέλεσμα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φυσικά, όταν μιλούμε για απόλυτη εναρμόνιση, μάλλον τίνουμε, γιατί αυτή είναι και η διατύπωση λίγο πολύ τη Επιτροπή, μάλλον τίνουμε προ τον κανονισμό παρά προ την οδηγία. Αλλά όπω είπα, για μένα μεγαλύτερη σημασία έχει το περιεχόμενο. Βάσει το περιεχομένου θα πρέπει να ε, κρίνουμε τι είδου νομοθέτημα θα ε, προταθεί. Ευχαριστώ για τη συνεργασία, ευχαριστώ όλους ε, τους συναδέλφους για την βοήθεια που μου προσέφεραν σε αυτή τη διαδικασία και στο επόμενο βήμα θα έχουμε βέβαια την συνοπτική κατάρτιση, τη συνοπτική ε, ενσωμάτωση των τροπολογιών στο κείμενο και αν θα επανέλθουμε. Κύριε Νετφέλτ, ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος με παρακάλεσε να τον αντικαταστήσω για περίπου μία ώρα και ε, καθώς έχω και την επόμενη έκθεση στην ημερήσια διάταξη θα συνεχίσω εγώ να μιλάω. Ταυτόχρονα όμως θα ε, ε επιβάλλω αυτοπιθαρχία στον εαυτό μου και θα μείνω πολύ σύντομη. Η επόμενη έκθεση λοιπόν έχει να κάνει με την αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικά επιτεύγματα και μελλοντικέ προκλήσεις. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας. 124 τροπολογίες. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω δηλαδή ότι προξενεί τόσο, ότι γεννά τόσο έντονο ενδιαφέρον στους συναδέλφους η έκθεση αυτή. Βλέπω ότι έχουν καλύψει με τις τροπολογίες τους ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, 224 τροπολογίες όπως είπαμε, και βλέπω ότι προσπαθούν να ενσωματώσουν τα θέματα σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα πρακτικά θέματα ε, ψηφίζουμε στις 15 ή 16, 15 νομίζω Ιουνίου, στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής μας και ε, στοχεύουμε για την ε, Ολομέλεια του Ιουλίου, εφόσον βέβαια έχουμε εγκαίρως τη μετάφραση των κειμένων. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπουμε προς το παρόν. Προφανώς τις 224 τροπολογίες θα προσπαθήσω να τις συμπτύξω σε πιο μικρό αριθμό. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα δώσει τη σχετική υπόσχεση, δεν τα κατάφερα όμως γιατί δεν πρόλαβα. Θα τα καταφέρω όμως με βεβαίω ότι θα βρω το χρόνο ώστε μέχρι την επόμενη συνεδρίαση ε, και μάλιστα εγκαίρω να έχουμε το χρόνο και να διαπραγματευτούμε και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Όπω είπα, καλύπτουν βέβαια το φάσμα θεμάτων οι τροπολογίε αυτέ. Γι' αυτό σκοπεύω να επικεντρωθώ μόνο σε ορισμένα από αυτά τα θέματα. Καταρχά, ενδιαφέρον είναι το ότι και ότι η έκθεση αφορά την αξιολόγηση τη αντιτρομοκρατική πολιτική, δηλαδή έχει αναδρομική έχει μάλλον στραμμένο το βρέμα προς τα πίσω ε, πολλοί είναι οι συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι κοιτάνε προς τα μπρος, προς το μέλλον και προσπαθούν να διαμορφώσουν τις πολιτικές για την καταπολέμηση τρομοκρατίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εν ώψη των μελλοντικών εξελίξεων. Αυτό δεν το κρίνω βέβαια ως ε, εσφαλμένο κατά ανάγκη, απλώς κατά την διατύπωση του καταλόγου και των υποδείξεών μου για τις ψηφοφορίες θα λάβω υπόψη το, τη διάσταση αυτή. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες στόχο έχουν να περιορίσουν το φάσμα, το πεδίο της αξιολόγησης. Αυτές θα τις υποστηρίξω. Η αδίποτε δημόσια πολιτική, ακόμη και η αντιτρομοκρατική πολιτική, θα πρέπει να είναι εκτεθειμένη σε έλεγχο διεξοδικό και αυτό είναι καθήκον δικό μας, δικό μας είναι καθήκον μας ως πολιτών να μπορούμε ε, και να προσπαθούμε να ελέγχουμε την εφαρμογή των πολιτικών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτη παρατήρηση. Πολλές από τις τροπολογίες σχετίζονται με τα δικαιώματα των θυμάτων Εδώ θα προσπαθήσω να πόσο συμβαστικέ προτάσει. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό το θέμα. Θα προσπαθήσω να τι ενσωματώσω έτσι ώστε να εγγραφούν μέσα στο πλαίσιο, στο πεδίο τη ε, προτάσεω, να βρουν τη θέση του. Αλλά είναι τόσο πολλέ οι προτάσει που θα προσπαθήσω να τι ομαδοποιήσω ώστε να μην γίνει και υπερβολικά μακροσκελή αυτή η έκθεση. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση για το κόστος της πολιτικής της αντιδρομοκρατικής. Οι σχετικές προτάσεις έχουν ε, ολοκληρωθεί, θα τις έχετε λάβει πιστεύω. Θα δείτε μια άτυπη παρουσίαση, μάλλον την 1η ε, Ιουνίου θα την οργανώσουμε, θα προσκαλέσουμε τους κοιόδης και τα λοιπά και όποιον είναι ενδιαφερόμενο. Πάντως γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουμε καμία ιδέα για το πόσα χαλάμε, πόσα δαπανάμε, δαπανούμε για την αντιτρομοκρατική μας πολιτική πράγμα το οποίο βεβαίως μας συγκλονίζει ο συμπέρασμα. Όπως επίσης και το γεγονός ότι είναι πολύ ασαφής η ιδέα που έχουμε ε, περί του οικονομικού φόρτου που επομίζονται οι επιχειρήσεις μας. Μαζί με το πόσα χαλάμε εμείς ε, για την τρομοκρατική πολιτική, πιστεύω ότι ε, θα έχουμε ένα πρώτο βήμα μάλλον, όχι βέβαια το τελευταίο, για την ανάλυση του συνολικού κόστους της αντιτρομοκρατικής πολιτικής. Επίσης, και νομίζω ότι αυτό καθίσατε και από τις τροπολογίες εφές, βλέπω ότι είναι αρκετή εκείνοι που αντιδρούν με επιχειρήματα αντίστοιχα με αυτά της Επιτροπής και του Συμβουλίου που λένε «Α, παρά είναι φιλόδοξη αυτοί οι...» ε, ε, πρόθεση, το εγχείρημα αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια ανάλυση λεπτομερή κτλ. Κοιτάξτε όμω, οι ΗΠΑ έχουν ε, τουναντίον αντίον ε, επιτύχει ένα πολύ υψηλό βαθμό λεπτομέρεια και ελέγχου του κόστου, και εφόσον μπορούν με διάφορε μάλιστα επιτροπέ και όργανα οι ΗΠΑ, οι Αμερικανοί δηλαδή να το κάνουν, γιατί όχι. Και μια και έχω ε, σύνδρομο σκυζοφρένειας και πολλαπλών προσωπικότητων, αλλάζω καπέλο και δίνω το λόγο στον κύριο Μπουσουτήλ ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε υπό την ιδιότητα που έχετε τώρα σαν Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και υπό την ιδιότητα σας ως ηγήτρια. Άκρος ε, ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Θα είμαι πολύ σύντομος. Εκπροσωπώ και την κυρία Χάνκης, εκπρόσωπο του ΕΛΚ, σκιώδη του ΕΛΚ, που μου ζήτησε να παρέμβω εκ μέρους της. Δύο βασικά θέματα τίθενται πάνω σε αυτά διαφωνεί σε κάποιο βαθμό το ΕΛΚ με την έκθεσή σας. Πρώτο σημείο, γιατί έχουμε μια πολιτική αντιτρομοκρατική εν πρώτης. Φαίνεστε να βασίζεστε επί της υποθέσεως ότι η πολιτική αντιτρομοκρατική οδηγεί σε παράνομη και υπερβολική συλλογή στοιχείων και παραβίαση κάποιων κανόνων και δικαιωμάτων. Το στο δεδομένο αυτό. Δεν θεωρούμε ότι αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα απαραίτητα. Προφανώς δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην οικονομική πτυχή της αντιτρομοκρατικής πολιτικής και διατείνεστε ότι το οικονομικό κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό, υπερβολικά υψηλό. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένα παράδοξο στην αξιολόγηση στρατηγικής αντιτρομοκρατικής. Ποιο είναι το παράδοξο. Δεν μπορεί να αξιολογήσει κανείς με βαθμό βεβαιότητας πόσες ζωές έχεις διασώσει. Άρα πόσο αποτελεσματική είναι η στρατηγική σου. Το ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό επακριβώς δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει κανείς μια αντιτρομοκρατική πολιτική διότι σώζονται ζωές σε αυτή την αίθουσα όλοι μας τα ασφαλείς όμως αυτό κοστίζει κάτι ε, χρειάζεται υπηρεσία ασφάλειας που μας προστατεύει και είμαστε ασφαλείς και δεν μας ανατινάζουν ποιο είναι το όφελος της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής εάν δεν μπορείς να δηλώνεις επακριβώς πόσες ζωές έχουν σωθεί. Η αξιολόγηση της αντιτρομοκρατικής ε, πολιτικής είναι δύσκολο να γίνει, πολύ δύσκολο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε μια αντιτρομοκρατική πολιτική και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμπεράνουμε απαραίτητα ότι είναι υπερβολικό το κόστος για κάτι τέτοιο αληθεύει και συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει και ένα κόστος και για τον τομέα και για τους άλλους εμπλεκομένους φορείς αλλά θα πρέπει να προσέξουμε μέχρι πού μπορούμε να προωθήσουμε να θέσουμε αυτό το επιχείρημα. Όπως είπατε υπάρχουν 224 τροπολογίες, τις εξετάσαμε. Θεωρούμε ότι βασικά είναι πολύ επικοδομητικές ε, τροπολογίες και προφανώς Περιμένουμε έναν καλό συμβιβασμό επί των τροπολογιών. Κάποιε τροπολογίες προφανώς είναι πολύ δύσκολο να τις δεχτούμε. Σας βλέπω που κουνάτε το κεφάλι σας και ελπίζω ότι τις επόμενες μέρες θα συζητήσουμε επικοδομητικά διότι έχουμε πάρα πολλά ισχυρά συναισθήματα για το θέμα και απόψει και την έκθεσή σα, και πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο να πετύχουμε ισχυρή πλειοψηφία για την έκθεση αυτή. το ότι υπάρχουν τόσες πολλές τροπολογίες αποδεικνύει ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική. Αποδεικνύει όμως ότι είναι και επίμαχη. Βασίζομαι σε εσά κυρία Πρόεδρε να μαζέψετε τους και και να καταλήξουμε όλοι μαζί σε μια ικανοποιητική συμβαστική λύση. Με ξέρετε. Εγώ έχω αυτό τον προσανατολισμό. Θέλω ε, συνένεση. Ο κύριος Δίες Δεμέρα έχει το λόγο. Bueno, Ευχαριστώ πρόεδρε και η συγγήτρια μαζί. Θα επαναλάβω αυτό που είπα πριν από 10 περίπου λεπτά. Το άρθρο 6 της Χάρτας των Θεμελιών Δικαιωμάτων αναφέρει την ασφάλεια ως θεμελιώδη αξία. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε επαρκή σημασία σε αυτή την έκθεση. Σίγουρα οι 224 τροπολογίες εκ των οποίων 38 είναι δικές μου ε, έχουν αυτό το στόχο ε, αλλά οφείλεται και στο γεγονός ότι πέντε επιτροπές νομοδοτούν για αυτό το ζήτημα οπότε ε, σίγουρα όλοι προσπαθούμε να είμαστε επικοδομητικοί εγώ ιδιαιτέρως αλλά καταλαβαίνετε γιατί υπάρχουν τόσες τροπολογίες. Εγώ στις 38 μου τροπολογίες ε, αναφέρομαι σε πέντε θέματα. Πρώτον, η τρομοκρατία αποτελεί πραγματική απειλή, πραγματική απειλή, δεν αποτελεί κατοσκεύασμα της διανόησης ούτε φαντασίωση. Δεύτερον, η τρομοκρατία θα πρέπει ε, να καταπολεμάται με δημοκρατικό τρόπο, χωρίς καμία αμφιβολία. Τρίτον, η τρομοκρατία ε, είναι διασπαστική τρομοκρατία, αναρχική τρομοκρατία, ε, ισλαμιστική τρομοκρατία ή τρομοκρατία των ε, βαρών των ναρκωτικών. Τέταρτον, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι δημοκρατικός αγώνας στον οποίο συμμετέχουν κυβερνήσεις και ιδιαίτερα οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέμπτον, οι διεθνείς διασυνδέσεις ανάμεσα σε τρομοκρατικές ομάδες και οργανωμένο έγκλημα. Μην ξεχνάμε τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Κολομβία, στη Γουατεμάλα. Προσέξτε τι είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας πολύ πρόσφατα, ο κύριος Άλβαρο Κολόν. Ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως συμβαίνει και στην Κολομβία, διότι αυτά που συμβαίνουν στην Κολομβία, στο Μεξικό και του Γατεμάλα είναι ότι το κράτος δεν μπορεί να φτάσει, δεν έχει πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της επικράτειάς του, διότι ε, βρίσκονται υπό τον έλεγχο των τρομοκρατών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη μεριά, έχουμε πρόβλημα επικάλυψης αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει να επαναβεβαιώσουμε το δημοκρατικό έλεγχο των μέσων που χρησιμοποιούνται εναντίον της τρομοκρατίας. Και αυτό είναι η αφετηρία. Το σημείο κίνησης. Ε, αλλά αυτό που είναι το βασικό, το πιο βασικό από όλα είναι η βοήθεια στα θύματα. Η βοήθεια στα θύματα θα πρέπει να είναι παντού και πάντοτε παρούσα. Αυτά είναι τα βασικά σημεία τα οποία ήθελα εγώ να θίξω. Όπως είπε ο κ. Μπουσούτιλ, ε, ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ευρεία συνένεση και θα είμαστε ε, ε, πολύ επικοδομητικοί. Ευχαριστώ. Okay, Καλώς. Ευχαριστώ. Βλέπω πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας και θα είμαι πιο αυστηρή. Σας παρακαλώ λοιπόν συνάδελφοι, αν μπορείτε να είστε λίγο πιο σύντομοι. Η κυρία Χέντιν υπομένει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστώ τη Σοφίντ Βέρτ, έξοχη δουλειά που έκανε. Σας και όδηση συγγήτρια, θα προσπαθήσω να εκφράσω την άποψή μας, αγγλιστή παρόλο που ήθελα να μιλήσω στα σουηδικά, Στόχος μας είναι μια ισορροπημένη έκθεση που θα καθορίζει μια αποτελεσματική αντιτρομοκρατική στρατηγική που σέβεται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πιστεύουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να είναι η πηξίδα για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ενώσης σε αυτόν τον τομέα και για τα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων. Η πρόληψη, ανείχνευση και η δίωξη των τρομοκρατών θα πρέπει να αποτελούν κομμάτι της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Συστημική στρατηγική χρειάζεται. Δεν θα πρέπει να βασίζεται επί καταστάσεων επιγουσών, αλλά επί στρατηγικής θα διαμορφώνεται βάσει αναγκών. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματική όσον αφορά το κόστος, να αποφεύγονται επικαλύψεις των μέτρων, των θεσμών και των διαφόρων υπηρεσιών. Υποστηρίζουμε αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση των τρομοκρατών αλλά θα πρέπει να διερευνήσουμε τους τρόπους. Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση. Πολλές τροπολογίες είναι αντιφατικές από αυτές υπευλήθησαν και δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι εμείς τι σημαίνει ένα πάνελ ανεξαρτήτων εμπειρογνωμών, Πρέπει να το συζητήσουμε και το διευκρινίσουμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Τέλος, όσον αφορά τα θύματα των τρομοκρατών πρέπει να κάνει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποβάλαμε σχετικέ τροπολογίες και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τροπολογίε που υπευλήθησαν από άλλα μέλη ε, στα πλαίσια συμβιβασμού. Ελπίζουμε να μην έχουμε τόσο πολλές τροπολογίες στο τέλος και ελπίζω ότι η έκθεση θα είναι καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Χιμένες έχει το λόγο. Eh, Είπατε ότι λάβατε πολλές ε, προτάσεις τροπολογιών και ότι θα εστιαστείτε στα πιο βασικά θέματα. Ε, θα ήθελα λίγο πιο συγκεκριμένα να μου πείτε ποια είναι αυτά τα βασικά θέματα στην καταπολέμηση τρομοκρατίας. Ε, εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι η κοινή ασφάλεια όλων των πολιτών, όσο και αν αυτό κοστίζει. Έχω υποβάλει πολλές τροπολογίες ε, που αφορούν πιο πολύ τα θύματα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είπατε ότι το ζήτημα των θυμάτων το θεωρείτε πολύ σημαντικό και ότι θα υποβάλλετε ε, συμβιβαστικέ τροπολογίε. Ελπίζω να μην είναι υπερβολικά απλουστευμένε, υπεραπλουστευμένε και να μπορώ να τι υποστηρίξω. Όταν μιλάμε για θύματα, υπάρχουν δύο τύποι θυμάτων. Τα πραγματικά θύματα, αυτά δηλαδή τα οποία ευλάθησαν, και τα ενδυνάμει θύματα τα οποία είμαστε όλοι εμείς, όλοι οι υπόλοιποι. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και τις δύο αυτές κατηγορίες θυμάτων και τα ενδυνάμει θύματα και δεν θα πρέπει να αφιστούμε προσπαθειών και κόστους. Και κυρίως να μην εφησυχάσουμε και πούμε ότι τώρα πια δεν έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ. Ε, μην ε, ε, ξεχνάμε ότι όποιοι ασχολούνται με αυτό το θέμα και μιλούν με άτομα που ασχολούνται με την καταπλέμηση τρομοκρατίας γνωρίζουν πολύ καλά πως σχέδια, τρομοκρατικά σχέδια υπάρχουν πάντοτε, συνεχώς. Συνεπώς ε, δεν θα ήθελα να μειώσουμε την ένταση του αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας. Ε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολλούς τύπους ε, τρομοκρατίας, όπως είπε ο κ. Διαθεμέρα, στον κυβερνοχώρο, ναρκοτρομοκρατία κλπ. Μην τα ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Κυρία Ζήπολ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να περιοριστώ σε δύο-τρία σημεία. Εάν δηλαδή χρειάζεται καταπολέμηση δημοκρατία, βεβαίω και χρειάζεται. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με το που βλέπουμε μια σφραγίδα καταπολέμηση τρομοκρατία να δεχόμαστε το κάθε τι. Όχι βεβαίω, γιατί και στην καταπολέμηση τρομοκρατία υπάρχουν διαφορετικά μέτρα, υπάρχουν μέτρα αποτελεσματικά, υπάρχουν μέτρα λιγότερο αποτελεσματικά. Υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό το συνοθήλευμα των ε, μέτρων κάποια τα οποία δεν είναι καν παραδεκτά. Και άρα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε αν όντω είναι αυτά τα μέτρα παραδεκτά ή και απαραίτητα. Και επίση τα μέτρα τα οποία ε, κάποια φορά μπορεί να αποφασίστηκαν για την καταπολέμηση τρομοκρατίας δεν είναι δεδομένο ότι πρόκειται να εξυπηρετήσουν σε κάποιον άλλον σκοπό. Φέρει πίνη αποθήκευση των δεδομένων. Είχαμε αποφασίσει με δεδομένο τον κίνδυνο τρομοκρατικών αποθέσεων επιθέσεων ε, την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, ενώ σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιήθηκαν ε, αποτελεσματικά, σε κάποια άλλα κράτη-μέλη η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά αυτά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά σε ε, άλλες λειτουργίε, εξυπηρέτησαν άλλου σκοπού, καθημερινή δηλαδή εγκληματικότητα, καταπολέμηση καθημερινή εγκληματικότητα, έτσι ώστε ε, τελικά καταστρατηγήθηκε ο λόγος για τον οποίο συλλέχθηκαν αυτά τα δεδομένα και βέβαια και το κόστος το οποίο εν τέλει σημαίνει αυτή η συλλογή και διατήρηση στοιχείων αστυνομικών αρχείων και το καθεξής. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη για να δούμε αν η αναλογικότητα ισχύει ή όχι. Τελευταίος ο κ. Άλμπεχτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον κύριο ε, Διασδεμέηρα, ο οποίο ε, μου ανέγνωσε το άρθρο 6 τη συνθήκη. Δεν το είχα υπόψη. Φυσικά θα ήθελα και να απαντήσω όμως ότι άλλο είναι να ε, βλέπουμε τα, τη διατύπωση αυτή της θεμελιώδους ελευθερίας, της, του δικαιώματος υπό το πρίσμα ενός δημοκρατικού και φιλελεύθερου κράτους, κρατικής δομής, και διαφορετικό αν το δούμε από το πρίσμα ενός αυταρχικού κράτους, το οποίο σαν στόχο έχει να περιορίσει μέσα από τις κρατικές δομές τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν μπορεί δηλαδή οι κρατικές δομές να βρίσκονται υπεράνω, να τίθενται υπεράνω των ίδιων των πολιτών. Εξαρτάται ως εκ τούτου από το για ποιο κράτος μιλάμε και για ποιες κρατικές δομές μιλάμε. Το ίδιο θα πρέπει να βλέπουμε πάντα όταν αναλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα ή επιλέγονται κάποιες ε, μέθοδοι. Δεν είναι πάντοτε κατάλληλα τα μέτρα σε κάθε κράτος. Άλλο το φιλελεύθερο και άλλο το κράτος το αστυνομικό, το κράτος της καταστολής. Αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη. Για τις παρατηρήσεις του κυρίου Μπουζούτσιλ. Θα ήθελα να επισημάνω, Σάιμον, ότι είναι κάπου, είμαι κάπως επιφυλακτικό, διότι εάν εν τέλει δεν υπάρχει ασφάλεια που να μας προστατεύει, εάν δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία να μας προστατεύουν, καθημερινά θα έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις. Αν δεν είχαμε εδώ την ασφάλεια στην είσοδο των ε, κτηρίων, θα μας είχαν την στον αέρα. Λες εσύ. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Ασφάλεια δεν είναι μόνο να περιορίζουμε τις ε, δραστηριότητες με την έννοια την αστυνομική. Ασφάλεια σημαίνει ταυτόχρονα και ουσιαστική απονομή δικαιοσύνη. Υπάρχει και μια καλή κοινωνική πολιτική που οδηγεί στην ασφάλεια, η, εξασφάλιση ενός βιωτικού επίπεδου ικανοποιητικού που να μην σπρώχνει, να μην οθεί τους ανθρώπους προς την ανάληψη τέτοιων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Και επίση θεωρώ ότι είναι απόλυτα θεμητό το να ζητούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο των μέτρων για την καταπολέμηση τρομοκρατία. Το έχουμε δει αυτό άλλωστε στην πράξη. Πολλά ήταν τα μέτρα στα τελευταία 5-15 χρόνια τα οποία εσύχθησαν για λόγου καταπολέμηση τρομοκρατία που όμω έπληταν άμεσα συγκεκριμένα άτομα και τι ε, ατομικέ του ελευθερίε ε, χωρί να προσφέρουν κάποιο ισοδύναμο επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Άρα, στο ερώτημα πώ θέλουμε να διαμορφωθούν στο μέλλον τα μέτρα για την καταπολέμηση τρομοκρατία, οι σχετικέ υπηρεσίε και τι είδους ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο θα ε, ορίσουμε για τι δραστηριότητε αυτέ, απάντηση δεν έχετε δώσει. Δεν μπορούμε τις πολιτικές ελευθερίες να τις υπαγάγουμε στην, ε, στο σκοπό της καταπολέμησης τρομοκρατίας. Επίσης, όταν ε, μιλούμε για τρομοκρατία υπάρχουν διαφορετικές ε, έννοιες, γιατί ακούγονται, ε, ακούγονται όροι όπως τρομοκρατία των βάρων των ναρκωτικών ή τρομοκρατία, κυβερνοτρομοκρατία του κυβερνοχώρου δηλαδή, ή ακόμη και τρομοκρατία των ε, αγωνιστών για τα δικαιώματα των ε, ζώων. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τον ε, βαθμό σοβαρότητας του κάθε φαινομένου και της τρομοκρατίας, της οργανωμένης, γιατί η τρομοκρατία ο, ο όρος, ο είδος της τρομοκρατίας είναι ασαφής. Η συμφωνία πλαίσιο για την τρομοκρατία που έχουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχει αποτελέσει πάντοτε την βάση για την ανάληψη, για τη λήψη αποφάσεων, είναι πια ξεπερασμένο και θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σαφή ορισμό τη τρομοκρατία με βάση τον οποίο θα ορίσουμε και την πολιτική μα. Δηλαδή, ποιο είναι ο στόχο τον οποίο τίνουμε. Να σταματήσω προς το παρόν εδώ με μία μόνο παρατήρηση, κλείνοντας για, τον, για την κυβερνοτρομοκρατία, ε, γιατί έχω υπόψη για τη δική μου τουλάχιστον εκλογική περιφέρεια ότι υπάρχουν ε, <laughs> υπάρχουν ε, μονάδες αστυνομίας, της οι οποίες είναι υποτίθεται εξειδικευμένες και ειδικά αφιερωμένε στον αγώνα για την καταπολέμηση της κυβεροτρομοκρατίας, αλλά τα κομπιούτερ τους δεν είναι καν συνδεδεμένα στο ίντερνετ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αποτελεσματική είναι η δράση τους. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εδώ τελείωσε ο κατάλογος των ομιλητών. Στον κύριο Σίφερ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω εδώ σημειώσει ότι ίσω θα να παρέμβει. Δεν έχετε σχόλιο. Καλώ. Έξοχα. Σας ευχαριστώ όλους σας πάρα πολύ. Θα απαντούσα στον κύριο Μπουσουτήλ, αλλά έπρεπε να αποχωρήσει το μεταξύ. Παρ' όλα αυτά θα το απαντήσω γενικότερα. Θα ήθελα να τον καθησυχάσω βεβαίως όπως και οποιοδήποτε άλλος αισθάνομαι ότι η τρομοκρατία θα πρέπει να καταπολεμηθεί αναμφισβήτητα. Κανείς σε αυτή την αίθουσα συνεδριάσεως ή στο Κοινοβούλιο θα αμφισβητούσε την ανάγκη που υπάρχει για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Νομίζω ότι προχωρά λίγο μακριά όταν υποθέτει ότι εγώ και άλλοι παριστάμενοι θα θεωρούσαν οδήποτε μέτρο αντιτρομοκρατικό να είναι παράνομο εισφαλμένο απλώς διότι θέτουμε κριτικά ερωτήματα. Υπάρχουν τα δύο άκρα. Είτε θεωρεί κανείς ότι οποιοδήποτε μέτρο αντιτρομοκρατικό είναι καλό και δεν θέτει ερωτήματα, είτε απορρίπτει όλα τα μέτρα απ' την άλλη. Κάπου στη μέση θα πρέπει να καταλήξουμε. Ναι, θέλουμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, αλλά με έναν τρόπο που να ταιριάζει με τις δημοκρατικές μας προδιαγραφές. Όλοι το λένε αυτό πάντα. Όταν όμως έρχεται η ώρα για να τίθενται ερωτήματα και να διεξάγεται έλεγχος, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Η κυρία Χιμένες έθεσε ένα βασικό ερώτημα. Ποια είναι η ουσία της αντιτρομοκρατίας. Τι καταπολεμούμε, τι πολεμούμε. Αυτομάτως πάντα υποθέτουμε ότι η αντιτρομοκρατία έχει σαν στόχο την διαφύλαξη ζώων. Θέλουμε να διασώσουμε ζωές να προστατεύσουμε τον κόσμο. Δίκιο έχει ο κύριος Δεμέρα. Είναι βασική ευθύνη αυτή των δημοσίων αρχών η προστασία του κόσμου. Όμως θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαφύλαξης της ζωής. Όπως είπε και η Ισπανική Προεδρία μπορούμε να καταπολεμήσουμε και την βία στα σπίτια. Θα σώσαμε πολλά περισσότερα, πολλέ περισσότερε ζωέ να το κάναμε αυτό. Θα μπορούσαμε να επενδύσουμε στην ιατρική έρευνα και να σώσουμε και άλλε ζωέ. Σκοπό όμω των τρομοκρατών, και αυτό είναι που του διαχωρίζει από τους απλούς δολοφόνους είναι ότι αυτοί θέλουν να καταστρέψουν τον ιστό τη Ελεύθερη Δημοκρατική Κοινωνία. Θέλουν να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου. Θέλουν να καταστρέψουν τις ελευθερίες μας, πολιτικές μας ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Και αυτό τους διαχωρίζει από τους απλούς δολοφόνους. Άρα έχουμε ένα διτό στόχο. Άρα είναι ακόμα πιο σημαντικό να ελέγχουμε εκ του σύνεγγυ τι αντιτρομοκρατικέ πολιτικέ. Διότι αν έχουμε αντιτρομοκρατικέ πολιτικέ που θέλουν να διασώσουν ζωέ, αλλά υπονομεύουμε άθελά μας τον δημοκρατικό μας ιστό, τότε παίζουμε το παιχνίδι εκείνο που θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τη σωστή προσέγγιση. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που συζητούμε. Δεύτερο σχόλιο. Πάνω σε κάτι που έθεσε η κυρία Ζήπερ. Πρέπει να ελέγξουμε τις πολιτικές τις αντιτρομοκρατικές, διότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν υιοθετηθεί μέτρα τα οποία μας τα πούλησαν σαν μέτρα αντιτρομοκρατικά, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για τελώς διαφορετικούς σκοπούς. Ίσως σωστούς σκοπούς, αλλά αυτό θα έπρεπε να έχει καταστεί σαφές. Και εδώ είναι που διαφωνώ με τον Σάιμον Μπουσοτήλ. Έλεγχος ή το να θέτουμε κριτικά ερωτήματα δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε κάτι. Σημαίνει ότι διεξάγεται ένας έλεγχος, ότι ελέγχεις, βλέπεις αν χρειάζονται τα μέτρα, πόσο αποτελεσματικά είναι, αν χρειάζονται περισσότερα, λιγότερα μέτρα, διαφορετικά μέτρα. Διαβεβαιώ την κυρία Χιμένεθ ότι δεν θα είναι υπεραπλουστευμένο ένα συμβαστικό κείμενο για τα θύματα. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να καταλήξουμε σε κάτι που θα εκφράζει αυτό που θέλετε να πείτε, αλλά πιο συνοπτικά από θα από το κείμενο που θα είχαμε αν συναθρίζαμε ως για το κόστος τώρα, κάτι που σχολίασε ο Σάιμον Μπουσετήλ. Δεν θα εκτελούσαμε τα κοινοβουλευτικά μας, τα δημοκρατικά μας καθήκοντα σαν βουλευτές, αν δεν θέταμε το ερώτημα πόσο κοστίζει. Αξιολογούμε και το κόστος της ε, πολιτικής για τη δημόσια υγεία, που και αυτή έχει στόχο τη διάσωση ζώων. Γιατί να μην το κάνουμε και εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι το κόστος είναι υπερβολικό. Απλώς θέλουμε να γνωρίζουμε ποιο είναι το κόστος, διότι δεν έχουμε ιδέα. Και είμαστε το μέσο οικονομικής κρίσεως. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι. Κάνουμε περικοπές στη δημόσια υγεία, στην παιδεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Ο κόσμος έχει κατέβει στους δρόμους της Μαδρίτης. Στην Ελλάδα ο κόσμος απεργεί, διαμαρτύρεται κατά των περικοπών του προπολογισμού και εμείς λέμε ότι δεν ενδιαφερόμεθα για το κόστος της αντιτρομοκρατικής δράσης. Εγώ το βρίσκω αυτό απαράδεκτο. Δεν λέω ότι θα πρέπει να ξοδέψουμε ευρώ παραπάνω ή λιγότερο, αλλά ότι σαν βουλευτές πρέπει να ρωτήσουμε πώς ξοδεύουμε. Είναι θέμα δημοκρατικού ελέγχου. Πολλά άλλα σχόλια έγιναν. κυρία Χέτ για το θέμα του πάνελ των ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, ενό πάνελ ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, δεν ξέρω περί τίνο πρόκειται. Ποια είναι η ουσία όμω. Η μόνη αξιολόγηση που, θα, που πετύχαμε μέχρι τώρα γινόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ να το πω τώρα, δηλαδή, σαν ο κυνηγό να γίνεται θηροφύλακα που λέει στα αγγλικά. Δηλαδή να αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την ίδια τη πολιτική. Δεν είναι κάτι αξιόπιστο αυτό χρειαζόμαστε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Θα βρούμε τη σωστή διατύπωση. Ακούστηκαν κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις, νομίζω, από την κυρία Χάνκης, που πρότεινε να έχουμε κάποιο συνδυασμό μεταξύ αξιολογήσεως πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, αξιολογήσεως από ισότιμους φορείς και διευρύνσεως της, του συστήματος αυτού του ελέγχου και τώρα για τον Σάιμον Μπουσετήλ έχω ένα άλλο σχόλιο που απουσιάζει ο Σάιμον. Θέλουμε πολύ ισχυρή πλειοψηφία την έκθεση. Ναι είναι η απάντηση. Διότι παρόλο που ξεκίνησε και ουσιαστικά είναι μια αξιολόγηση, άρα κοιτάζουμε τι έγινε τελευταία δεκαετία, προφανώς θα εμπεριέχει και σημαντικές συστάσεις για μελλοντική αντιτρομοκρατική πολιτική, πολιτικές, άρα πρέπει να γίνει τώρα μια αποτίμηση, είναι σημαντική στιγμή, οπότε και εγώ με όλες τις πολιτικές ομάδες προσπαθήσω να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη για, το, για την έκθεση αυτή. Λοιπόν, αλλάζω ιδιότητα εκ νέου και επόμενο σημείο. Είναι το σημείο 7 που έχουμε στη μεστήριση είναι, είναι δίκτυο για ε, προειδοποίηση και κρίσιμε υποδομέ, δίκτυο συναγερμού και πληροφόρηση για τι κρίσιμε υποδομέ. Ο κύριο Λούχαν ε, είναι εισηγητή του ΕΛΚ. Μου ζήτησα να προεδρεύσω την τελευταία στιγμή. Δώστε μου μερικά λεπτά να ρίξω μια ματιά. Μάλιστα. Θα καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει τη δική μας Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της πιλωτικής φάσεως αυτού του δικτύου συναγερμού και πληροφόρηση της κρίσιμες υποδομές, το CWIN όπως είναι γνωστό, και άλλα βήματα που θα πρέπει να γίνουν. Θα καλέσω τον κύριο Heymans της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει μια εισαγωγή και μετά θα ζητήσω από τον εισηγητή να παρέμβει και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Λοιπόν, ο κ. Χάιμανς έχει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Με τα χαρά να σα παρουσιάσω ποιε είναι, ποιες είναι οι πιο πρόσφατε εξελίξει, τι πρόοδο πετύχαμε όσον αφορά την ανάπτυξη αυτού του δικτύου συναγερμού και πληροφόρηση για τι κρίσιμε υποδομέ. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το σύστημα αποτελούσε ένα τμήμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την ε, προστασία και τις κρίσιμες υποδομές. Ε, ξεκινήσαμε από το 2006 και σε αυτή τη φάση θέλαμε να έχουμε ένα σημαντικό εργαλείο για ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, για ανταλλαγή πληροφοριών και σύστημα συναγερμού για τα κράτη-μέλη σε περίπτωση επιθέσεως επικρισίμων υποδομών, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, και το σύστημα θα υποστήριζε και την εφαρμογή της οδηγίας για τον καθορισμό των ευρωπαϊκών κρισίμων υποδομών που θεσπίστηκε το Δεκέμβριο του 2008. Τώρα, μετά το 2006 έγινε μια μελέτη, ξεκίνησε μια μελέτη. Έγινε μεγάλη διαβούλευση με τα κράτη-μέλη περί του συστήματο, τι θα έπρεπε να κάνει το σύστημα και από αυτή τη βάση, ποια θα ήταν νομική βάση για το σύστημα. Προτάθηκε αυτή το Σεπτέμβριο του 2008 και μετά ξεκίνησαν συζητήσει όσον αφορά τη νομική βάση στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο αμέσως ξεκαθάρισε δύο πράγματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, βασικά τα κράτη-μέλη είπαν ότι μπορούμε να συζητήσουμε την νομική βάση για την πρόταση αυτή μόνο αν εξετάσουμε προσεκτικά το σύστημα. Θέλουμε να ξέρουμε περί τίνο πρόκειται, τι μπορεί να κάνει, πώ λειτουργεί κλπ. πριν να μπορέσουμε να συζητήσουμε τη νομική βάση. Το δεύτερο βασικό σημείο που απέρευσε από τι αρχικέ συζητήσει ήταν ότι τα κράτη-μέλη είπαν ότι δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα σύστημα συναγερμού Υπάρχουν ήδη αρκετά συστήματα συναγερμού στους διάφορους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα προστασίας των κρισίμων υποδομών και αυτές οι τομαϊκές προσεγγίσεις ε, προτιμούνται από τα κράτη-μέλη εν συγκρίση με την πρόταση που κάναμε εμείς να έχουμε ένα σύστημα που θα είναι διατομεακό ε, για την προστασία των κρισίμων υποδομών. Εμείς τι είπαμε. Αν τα κράτη-μέλη θέλουν να εξετάσουν το σύστημα, καλώς. Θα αναπτύξουμε το σύστημα σε πιλωτική φάση για να το δουν πρώτα. Αυτό κάναμε. Για να το δουν τα κράτη-μέλη, να παίξουν μαζί του, να δουν κατά πόσο αποκρίνει τι απαιτήσει του και να προτείνουν κάποιε περαιτέρω αλλαγέ και βελτιώσει που θα μπορούσαμε να επιφέρουμε στο σύστημα, ώστε να ανταποκρίνει τι απαιτήσει των κρατών μελών. Επίση, για να εξασφαλίσουμε την σωστή ανταλλαγή απόψε στα κάτι μελη διοργανώσαμε αξιολόγηση τη πιλωτική φάσεω, κάτι που έγινε πέρσι το πιλωτικό σύστημα διατέθη στα κράτη-μέλη τον Απρίλιο του 2010 και ολοκληρώθηκε η εξολογήση του συστήματος τον Οκτώβριο και τα αποτελέσματα, τα πορίσματα της εξολογήσεως δόθηκαν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, οπότε μπορέσατε να δείτε ε, ποια ήταν τα διάφορα σχόλια και οι παρατηρήσεις. Η εξολόγηση του συστήματος συζητήθηκε μετά με τα κράτη-μέλη στα σημεία συνεδρίαση των σημείων επαφής εκείνων που ασχολούνται στα κάτι μέλη με, τα, με την προστασία των υποδομών συνεδριάζουν και τι απέρευσε. Ότι γενικά υπήρχε υποστήριξη για το σύστημα, αλλά θεωρήθηκε επίση ότι χρειάζεται και άλλε βελτιώσει. Βασικό συμπέρασμα ήταν ότι το σύστημα προσέφερε καλύτερη λειτουργικότητα, περισσότερη λειτουργικότητα από ό,τι χρειαζόταν, άρα ήταν λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι χρειαζόταν για κάποιου εμπειρογνώμονε τουλάχιστον των κρατών μελών και κάποια άλλα σημεία απέρευσαν. Σύντομη περίοδο υπήρξε τη χρήση του συστήματο, περίπου έξι μήνες μόνο πριν γίνει αξιολόγηση. Δεν είχε γίνει εκπαίδευση όλα τα κατημέλη, όμως το συμπέρασμα ήταν ότι πετύχαινε το στόχο το σύστημα. Και αναγνώρισαν τα κράτη-μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα. Αυτό είπαν τα κράτη-μέλη. Θα είδατε από την έκθεση ότι δεν υπήρχε συμφωνία επί δύο βασικών ζητημάτων που είχαν τεθεί ευθύ εξ αρχή. Πρώτον, κατά πόσο το σύστημα θα μπορούσε να εξετάζει διαβαθμισμένες, περιορισμένες πληροφορίες των κρατών μέλων. ήταν διαρρεμένα τα κάτι μέλη 50-50. Κάποιοι έλεγαν ότι κάποιες από τις εκθέσει εκθέσεις που υπάρχουν και αφορούν το πώς ευάλωτες είναι οι κρίσιμες υποδομές είναι σημαντικές εκθέσεις και το σύστημα θα έπρεπε να επιτρέπει την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών και με άλλα κράτη-μέλη. Η άλλη πλευρά έλεγε ότι πρέπει να διαβρύνουμε τη χρήση του συστήματος και να διατεθεί και στους α, εκείνους που, τους φορείς των κρισίμων υποδομών, ούτω ώστε να μπορούν να βλέπουν τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται από τους χρήστες του συστήματος και τελικά κατέστη ανέφικτο να συμφιλειωθούν οι δύο διαφορετικές ε, θέσεις. Συμπέρασμα. Να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανάψει του συστήματος να βελτιώσει την χρήση αυτού, να γίνει απλούστερο και να οργανωθεί εργαστήριο με τα κρατημέλη για περαιτέρω συζήτηση των βελτιώσεων. Το εργαστήριο έγινε, πραγματοποιήθηκε φέτος στις 17 Μαρτίου. Επειδή δεν υπήρχε συμφωνία όσον αφορά τις διαβαθμισμένες πληροφορίες, εμπιστευτικές πληροφορίες, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση άνευ περαιτέρω συζητήσεων με τα κρατημέλη. Επ' αυτής της Ενημερώσαμε τον Επίτροπο, την Επίτροπο. Συμφώνησε με τα συμπεράσματα συνεδριάσεως. Αποφάσισε από την πιλωτική φάση να προχωρήσουμε. Την πιλωτική φάση που ξεκίνησε από πέρσι τον Απρίλιο να πάμε στο πλήρες σύστημα, στην παραγωγή, στη φάση παραγωγής. Και οι αλλαγέ που απορρέουν από την αξιολόγηση αποφάσισε Επίτροπο ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν και θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα να έχει το σύστημα αυτόματης μετάφρασης για το θέμα των διαβαθμισμένων πληροφοριών το αφήνουμε για την ώρα μέχρι ότου κουβεντιάσουμε περαιτέρω με τα κράτη-μέλη. Άλλο σημαντικό στοιχείο. Θα διπλασιαζόταν το κόστο του συστήματο αν ακολουθούσαμε, αυτή την ε, προσέγγιση όσον αφορά τι διαβαθμισμένε πληροφορίε, Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρόταση για τη νομική βάση για το σύστημα θα μπορούσε να αποσυρθεί. Η νομική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα έδωσε σχετική γνωμοδότηση χρειαζόμαστε μια νομική βάση για τέτοιο σύστημα αν πληρούνται μία από τις τρεις προϋποθέσεις. Πρώτη, η χρήση να είναι υποχρεωτική του συστήματος. Αυτό το συζητάμε τα κράτη-μέλη, το συζητήσαμε. Δεν υποστήριξαν κάτι τέτοιο τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, αν το σύστημα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπω το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εξετάζονται μη προσωπικά στοιχεία στο σύστημα. Και τρίτον, αν το σύστημα θα ε, επεξεργαζόταν ε, διαβαθμισμένες πληροφορίες. Εφόσον δεν πληρούνται αυτές οι συνθήκες, αποφάσισε ο Επίτροπος ότι θα αποσυρθεί η πρόταση αυτή για την νομική βάση και άλλη πρόταση για άλλη νομική βάση θα υποβληθεί αν πληρωθούν κάποτε κάποιες από αυτές, από αυτές τις συνθήκες. Εάν τελικά το σύστημα εξετάζει εμπιστευτικές πληροφορίες, αν συμφωνήσουν αυτόν το κάτι μέλη, τότε θα πρέπει να προβλέπεται νομική βάση. Ολοκληρώθηκαν σχεδόν οι διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις για την εφαρμογή των αλλαγών που ζητήθηκαν. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα ολοκληρωθεί το, σύμβαση και θα ξεκινήσει το σύστημα πριν το καλοκαίρι. Και το σύστημα μέχρι τέλος το έτος θα διατεθεί σε πλήρη λειτουργία για τα κάτι μέλη. Και μέχρι τότε μπορεί να συνεχιστεί η χρήση του πιλωτικού συστήματος. Αυτά είχα να πω εν είδη εισαγωγής και Ευχαριστώ ο κ. Λούχαν, ο συγκητή, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτέλους αρχίζουμε να συζητάμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας. Υπάρχουν πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα και πολύ άγνωστοι παράγοντες. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν για την παρουσίασή τη Ήταν πολύ λεπτομερής και χρήσιμη. Όπως είπε η Κομισιόν, ήδη υπάρχει ένα ιστορικό που ξεκινά από το 2005. Από τότε μιλούμε για τις ε, κρίσιμε υποδομέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κάθε φορά, κατά για κάποιο λόγο, αναβάλουμε τη συζήτηση. Κατά την άποψή μου αυτοί οι λόγοι δεν είναι βάσιμοι. Το καλό είναι ότι έχουμε πλέον την ε, ευκαιρία να το συζητήσουμε. Μετά από τόσα χρόνια διαθέτουμε πλέον ένα δίκτυο συνεργασμού και πληροφόρησης σε δύο πεδία. Ανεξαρτήτως όμως του, του, του τομέα του πεδίου, ε, αν είναι υγεία, μεταφορές, ε, τρόφιμα, εκπαίδευση ή οτιδήποτε άλλο, όλοι αυτοί οι τομείς, όσοι και αν είναι, θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να συζητούμε άλλες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε μιλήσει μόνο για τις τεχνικές πτυχέ. Τι θα κάνουμε με τα δεδομένα, πώς θα τα συλλέξουμε, πώς θα τα αποθηκεύσουμε, πώς θα εξασφαλίσουμε την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων κλπ. Όμως αυτά δεν είναι αρκετά. Ως πολιτικοί θα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη προσέγγιση. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω. η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού δικτύου συναγερμού και πληροφόρηση σε όλους τους ε, τομείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, είναι πάρα πολύ ε, ε, σημαντική. Τώρα θα εξετάσουμε το κατά πόσον θα συμπεριλάβουμε όλους τους τομείς στο ίδιο project, όπως λέει η Κομισιόν, ή αν θα πρέπει να ξεχωρίσουμε. Όμως θα πρέπει τα δίκτυα συναγερμού και πληροφόρησης να συνεργάζονται μεταξύ τους. Μόνο έτσι μπορούμε να ακολουθήσουμε αποτελεσματικές πολιτικές για όλους τους τομείς που είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελέγχθη ότι το 2008 υπήρχε, είχε γίνει μια πρόταση για την νομική βάση κατόπιν ανάλυσης. Ε, μόνο εν μέρη συμφωνώ με αυτό που είπε η Κομισιόν. Τα περισσότερα κρατημέλη συμφωνούν με την ύπαρξη νομικής βάσης. Και έχω και συγκεκριμένα νούμερα. 65,8% Ε, των, απαντήσεων ε, ήταν θετικές για την ε, θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Δικτύου Συναγερμού. 14 κράτη-μέλη είπαν ότι το σύστημα των δύο συστημάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα δύο συστήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διευρυνθούν και να βελτιωθούν. Σε ό,τι αφορά την γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην οποία αναφέρθηκε η Κομισιόν, να σας πω ότι δεν έχουν δοθεί οι σωστές πληροφορίες στα κράτη-μέλη. Το ερώτημα είναι, τα κράτη-μέλη συζήτησαν για αυτό το σύστημα μετά από πραγματική και εις βάθος ανάλυση ή όχι. Νομίζω ότι αυτό δεν συνέβη. Αυτή η ανάλυση δηλαδή δεν έλαβε χώρο σε όλα τα κράτη-μέλη. Έξι μήνες δεν λαβει χωρο σε ολα τα αρκετό χρόνος για να απαιτήσουμε μια συγκεκριμένη απάντηση. Άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω σήμερα είναι το εξή. Η απόσυρση της νομοθετικής πρότασης και η υποβολή καινούριας νομοθετικής πρότασης μου δημιουργεί ένα ερωτηματικό. Μήπως πρόκειται πάλι για στρατηγική αναβολής. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα αν θέλουμε να μιλάμε για ένα αποτελεσματικό σύστημα. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, θα πρέπει να κάνουμε βήματα, ε, συγκεκριμένα βήματα. Αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι ε, ως τώρα ε, είχαμε βάλει το θέμα κάτω από το χαλί. Θα πρέπει στο τέλος της συζήτησης να εκδώσουμε μια γνωμοδότηση ό,τι αφορά, να, μάλλον να πάρουμε θέση σε ό,τι αφορά το αν θα χρησιμοποιηθεί η νομοθετική πρόταση που υπάρχει ή αν θα εκδοθεί καινούργια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα άτομο έχει ζητήσει το λόγο. Η κυρία Μποσκούρτ. Θέλει κανεί άλλο το λόγο, μήπω. Κυρία Μποσκούρτ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πρώτη συζήτηση αυτού του θέματος. Έχω μία ερώτηση. Αν δούμε το θέμα της αξιολόγησης. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν λάβει ε, μέρος στην, στην ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, υπάρχει ενδεχομένως ένα θέμα ασφάλειας ε, στην ανταλλαγή αυτών των δεδομένων. Ίσως το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκές. Δηλαδή ε, θα έπρεπε η ανταλλαγή αυτή να γίνεται με ασφαλή τρόπο. Συνεπώς η ερώτησή μου είναι η εξής. Πότε θα αρχίσουν τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες, τι προσδοκούν και τι περιμένει η Κομισιόν Ο στόχο είναι να βασιστούμε σε εμπειρία που έχει αποκτηθεί από άλλα δίκτυα όπως το SIS, για παράδειγμα, το σύστημα πληροφοριών Schengen. Η Κομισιόν πότε θα επιταχύνει την ανταλλαγή αυτή, γιατί τελικά αυτός είναι ο στόχος, η αλλοενημέρωση. Αυτό είναι η προστιθέμενη αξία του συστήματος. Θα μπορούσατε να μας απαντήσετε σε αυτό το ζήτημα. Κομισιόν. Πώς λειτουργεί το σύστημα της ανταλλαγής πληροφοριών, πώς θα λειτουργεί όταν έχουμε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις. Είναι το σύστημα έτοιμο για αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια ιδέα για το πώς θα καθυστερήσουμε. Και μετά, Δύο ακόμα ερωτήσεις που πηγάζουν από αυτά που είπατε. Είπατε παρενθετικά για ε, μια ελεπικάλυψη και δεν κατάλαβα πολύ καλά τι ακριβώς εννοούσατε. Μήπως θα μπορούσατε να μου το διευκρινίσετε. Και μετά για όλο το, για το συνολικό project είπατε ότι θέλετε μέχρι το τέλος του 2011 να λειτουργεί όλο το σύστημα. Ε, όμως αυτή τη στιγμή κάποια κράτη-μέλη εξουσιάζουν ακόμα δισταγμούς. Πώς θα τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Ευχαριστώ. Εάν δεν θέλει να λάβει το λόγο κανείς άλλος συνάδελφος, αν συμφωνεί. Και μπορούμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή εν συντομία να δώσει απάντηση στις ερωτήσεις, κύριε Χέμανς. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δώσω τις απαντήσεις. Πάντως ε, είναι περιορισμένο αυτή τη στιγμή το σύστημα, αλλά μόνο στο πιλωτικό επίπεδο και σκοπεύουμε να το καλύψουμε να το επεκτείνουμε έτσι ώστε να καλύπτει όλου αυτού του διαφορετικού τομεί από τα κράτη-μέλη. Και ήθελα να υπογραμμίσω επίση ότι προφανώ δεν υπάρχει καμιά πρόθεση από πλευρό μα να αποκρύψουμε πληροφορίε. Πάντοτε πιστεύω δύναμε πρόθυμα ε, τις πληροφορίες που έχει αισθήσει η Επιτροπή σας. Και η συνεργασία μας αυτή ε, έχει την ίδια ε, διαφάνεια και σχέσεις με τα κράτη-μέλη. Αυτό βλέπετε και από την έκθεση ότι συμμετέχουν σε κάθε στάδιο επεξεργασίας και ανάπτυξη του συστήματος όπως και στην αξιολόγησή του. Η απόφαση για την νομική βάση προφανώς δεν έχει σαν στόχο να καθυστερήσει την εφαρμογή, την υλοποίηση του συστήματος. Από την εμπειρία όμως που έχουμε από τις διαπραγματεύσεις μας με τα κράτη-μέλη, θεωρήσαμε ότι αυτή είναι και η σωστή προσέγγιση και μας επέτρεπε και να ε, θεσπίσουμε ή να θέσουμε σε λειτουργία καλύτερα το ταχύτερο δυνατό το σύστημα, ώστε να μην, να χρειαστεί να περιμένουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο επίπεδο Συμβουλίου. Το γεγονό ότι δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει στο σύστημα όλα τα κράτη-μέλη βεβαίω αποτελεί επιλογή των ίδιων των κρατών μελών. Εμεί του έχουμε προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβαση στο σύστημα, εάν δεν προτιμούν δεν είναι υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιήσουν, αλλά φυσικά θεωρούμε ότι όσο πιο πολλά είναι τα κράτη-μέλη που το χρησιμοποιούν, τόσο πιο πολλά κράτη-μέλη θα αναγνωρίσουν και την προσθέμενη αξία προσφέρει αυτό και και τούτου θα προσελκυστούν ε, να το χρησιμοποιήσουν και άλλα κράτη-μέλη από την αξιολόγηση ωστόσο θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα σου προς την ασφάλεια. Είναι ασφαλές το σύστημα, όσο ασφαλές μπορεί να είναι οποιοδήποτε σύστημα σε σχέση με την εισαγωγή κωδικών πρόσβασης κτλ. Δεν έχουμε προβλήματα ως προς το απόρριτο, τουλάχιστον από τα κράτη-μέλη δεν μας έχουν δώσει τέτοιες ε, πληροφορίες. Για να σας διευκρινίσω και σχετικά με τις ε, ε, προτεραιότητες μας, με τις προσδοκίες μας. Εμείς σκοπεύουμε τώρα να προχωρήσουμε σε υλοποίηση αλλαγών με βάση τις παρατηρήσεις και των κρατών μελών που θα εισαχθούν εν, ε, στην ε, υπό το ισχύον σύστημα, υπό την ισχύουσα σύμβαση καλύτερα, ενώ τα υπόλοιπε παρατηρήσεις στην επόμενη. Οποιοδήποτε ζήτημα πάντως έχει σημανθεί θα αντιμετωπιστεί. Η ΙΣΠΑ στο κοινό κέντρο έρευνας υποδέχεται το σύστημα αυτό, είναι ο host δηλαδή για το σύστημα αυτό, δεν χρειάζεται μεγάλη υποδομή, ε, δεν είναι σύστημα δηλαδή ευρεία κλίμακα που να χρειάζεται περισσότερο εκτεταμένε υποδομέ και άρα θεωρούμε ότι θα συνεχίσει να το ε, ε, φιλοξενεί η ΙΣΠΑ με το Κοινό Κέντρο Ελέγχου. Το σύστημα επιτρέπει ταχύτατη διάδοση πληροφοριών με πολύ καλές περιόδου αντίδραση κάτω από ένα δευτερόλεπτο, όπως δηλαδή αναμένεται από ένα τέτοιο σύστημα. Πολύ ικανοποιητική η περίοδος ανταπόκρισης. Και θέλω να πω επίσης ότι εάν θέλει κανείς να προσαρμόσει το σύστημα έτσι ώστε να καλύπτει και ενδεχομένως απόρριτα ή με περιορισμένη πρόσβαση δεδομένα. Αυτό σημαίνει προσαρμογές όχι μόνο στο δικό μας επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών, δηλαδή επιπλέον κόστος ε, του όλου συστήματος, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι θα διπλασιαστεί το συνολικό κόστος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Και τώρα ας ακούσουμε τον κύριο Λούχαν, τον συνάδελφο για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις σας εύστοχες και ευπρόζεκτες. Θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ύπαρξη ενός νομοθετικού πλαισίου και ενός συστήματος, ε, ενός δικτύου συναγερμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μετά θα περάσω στο τι προτείνω ε, σε σχέση με τα δεδομένα, πώς μπορούμε να τα μεταχειριζόμαστε, τι είδους διαβάθμιση θα γίνεται, ποιος θα έχει πρόσβαση στη διαβάθμιση, ποια κράτη-μέλη και το καθεξής. Ε, βεβαίως αναμένω και περαιτέρω τροπολογίες όπως και συζητήσει στην υπόθεση αυτή, αλλά ας ξεκινήσω με ένα ερώτημα που απευθύνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι το εξή. Θα μπορούσατε να μας ορίσετε μια προθεσμία για το πότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ένα τέτοιο δίκτυο συναγερμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί χρειάζεται κατεπηγόντως. Και θέλουμε να το δούμε το ταχύτερο δυνατό σε εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επίσης, τα κράτη-μέλη εν μέρη μόνο μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ε, διαβουλεύσεις. Ε, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στις ε, διαβουλεύσεις πριν ληφθεί κάποια απόφαση. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να υποχρεωθεί να ε, λάβει μέρος σε ένα τέτοιο σύστημα, σε ένα τέτοιο δίκτυο. Αλλά το δίκτυο πρέπει να υπάρξει και να θεσπιστεί και να λειτουργήσει. Η Επιτροπή μας λέει τώρα ότι προτιμάει μια συλλογική προσέγγιση. Ε, πρόκειται για, μια... για ένα θέμα συζήτησης, το οποίο φαντάζομαι θα μας απασχολήσει και σε μια από τις προσεχείς ε, συνεδριάσεις. Θα πρέπει να αποφασίσουμε βέβαια σε ποιο βαθμό είναι δυνατή αυτή η προσέγγιση, αλλά και εφικτή οικονομικά. για δε τα διαβαθμισμένα δεδομένα. Πιστεύω ότι θα πρέπει και οι Υπουργοί των, Εσωτερικών και των Εξωτερικών, όπως και αυτοί, ε, και τα, όπως και τα Υπουργεία, ε, τα αρμόδια για την προσέγγιση των προσωπικών δεδομένων, ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη διαδικασία. Και θεωρώ ότι θα πρέπει η Επιτροπή να προσεγγίσει κατά τη διάρκεια της διαβουλεύσεως αυτά ακριβώς τα Υπουργεία. Πάντω ήθελα προς το παρόν όλοι οι συνάδελφοι να διαβάσουν την έκθεση ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να εκφράσω την ελπίδα την προσεχή φορά να γίνει μια ε, συζήτηση λεπτομερής. Και να έχουμε το ταχύτερο δυνατό το χρονοδιάγραμμα που έχω στήσει από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα ήθελε η Επιτροπή να απαντήσει. Κύριε Χέιβαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή δεν σκοπεύει να καταθέσει νέα νομοθετική πρόταση. Όπω εξήγησα και νωρίτερα, αποφασίσαμε να αποσύρουμε την νομοθετική πρόταση και μόνο εάν παρατηρηθούν περαιτέρω εξελίξεις, δηλαδή διατυπώσουν προς τώρα κράτη-μέλη την ε, επιθυμία να αναπτυχθεί ένα τέτοιο δίκτυο και κυρίως την επέκτασή του ε, για να περιλάβει και διαβαθμισμένα δεδομένα, τότε μόνο θα επανέλθει η Επιτροπή με νέα πρόταση. Προς το παρόν όμως η κατάσταση είναι αυτή και δεν σκοπεύουμε να καταθέσουμε νέα πρόταση. Ευχαριστώ, λίγο Με ναι, αυτό μπορούμε να καταλήξουμε. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια του κύριου Λουχάν. Συμφωνείτε από ό,τι βλέπω. Και πάμε στο επόμενο σημείο που είναι το υπαριθμό 8. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. ΕΝΙΣΑ. Αρμόδια για το, επί της ουσίας για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή Ήτρε με τον κύριο Τσίτσαστερ. Εμείς έχουμε αναλάβει μια γνωμοδότηση ε, που έχει αναλάβει ο κύριος Αλεξάνδρ Άλβαρο, συντάκτης γνωμοδοτήσεως, αλλά ας ακούσουμε πρώτα την πρόταση της Επιτροπής, την παρουσίαση για την αναδιατύπωση του κανονισμού που στόχο έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις σχετικές με την αναθεώρηση της εντολής της ε, αποκεντρωμένης υπηρεσία. Ο κύριος Άλβαρο. The point is that we've been reported... Από ό,τι μας λένε, η Επιτροπή, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δεν έχει έρθει ακόμη στην αίθουσα έπρεπε να είναι εδώ στις 10 και 25, σε 10 λεπτά. Ε, τότε ας ακούσουμε τον κύριο Άλβαρο. Και μετά την Επιτροπή. Για να μην ε, χάσουμε περισσότερο χρόνο. Μην ξεχνάμε ότι στις 12.30 θα έρθει η Επίτροπος Μάλστρομ. Και πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί με το χρόνο. Κύριε Άλβαρο, θέλετε να κάνετε την παρουσίαση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εάν περιμένετε ότι θα μιλάω επί 10 λεπτά μέχρι να έρθει ο πρόεδρος της Επιτροπής, τι να σας πω δεν έχω τόσο πολλά να πω και είναι πολύ συνεργαστικό το θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει αναλάβει επί της ουσίας η Επιτροπή Μηχανίας. Εμείς έχουμε γνωμοδότηση. Έχει φυσικά να κάνει με τις πτυχές ε, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων η δική μας γνωμοδότηση. Η συζήτηση για το ΕΝΙΣΑ λίγο πολύ έχει καλυφθεί στη γενικότερη συζήτηση στη σχετική με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Έχει το, τη σχετική πρόβλεψη για τον ε, προϋπολογισμό, έχει και την έδρα η οποία ως γνωστόν είναι ένας πολύ ωραίος ε, τόπος παραφερισμού, δεν ξέρω πόσο σκόπιμη είναι η επιλογή αυτή για σοβαρή δουλειά, η Κρήτη δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει όμως η Επιτροπή Βιομηχανίας όπως και εμείς πιστεύω έχει λίγο πολύ ε, συζητήσει θέματα σχετικά με την έδρα με την Ελλάδα που υποδέχεται την ενίσα ε, ίσως κάποια πράγματα, κάποιες διαφορετικές προτάσεις να ε, ε, τύχουν επεξεργασία στο μέλλον. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την κυβερνοτρομοκρατία, την κυβερνοασφάλεια, το κυβερνοέγκλημα και άλλα κυβερνοπράγματα. Και Δεν ξέρω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτσι επιφυλακτική ως προς την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Ο κύριος Λουαν μίλησε για κρισίμες ε, υποδομές. Στη δική του έκθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι διαβάζουμε σκοπεύει να αναπτύξει και μια μονάδα κυβερνοάμυνας και πέραν αυτή έχουμε και το ΕΝΙΣΑ. Ε, ερωτώ λοιπόν ε, πόσο αποτελεσματικοί μπορούμε να είμαστε εάν έχουμε τόσο μεγάλο κατακαιρματισμό των εργασιών μας. Θα ήταν σκόπιμο μάλλον ε, υπό, ε, υπό μια μεγάλη και κοινή ομπρέλα να υπαγάγουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες ε, κυβερνοασφάλειας. Θα δούμε βέβαια και με βάση την έκθεση τι μπορούμε να επισημάνουμε εμείς, διότι όπως είπα δεν έχει ακόμα κατευθεί το σχέδιο της εκθέσεως από την αρμόδια επιτουσίας επιτροπή. Έχουμε και την ε, η προθεσμία της 19ης Ιουνίου, για την οποία έχει προβλεφθεί να καταθέσει ο κύριος του τη του έκθεση Επιτροπή Βιομηχανίας, όπως και εμείς, και έχουμε τροπολογίες μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου από ό,τι φαίνεται για τη δική μας ε, γνωμοδότηση. Άρα ο καθένας μπορεί ήρεμα στις διακοπές του να σκεφτεί τι είδου τροπολογίες θέλει να καταθέσει στην έκθεση, στην, στο σχέδιο της γνωμοδότηση. Απλώς σχετικά με την κυβερνοεγκληματικότητα ε, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να προσφέρει επιπλέον η Ενίσα, τι είδου διάρκεια θα έχει η θητεία τη και ποιο θα είναι ο ρόλος του λεγόμενου Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται. Από τα τελευταία έγγραφα του Συμβουλίου υπάρχουν από ό,τι φαίνεται κάποια εκρεμή ζητήματα τα οποία πρόκειται να επεξεργαστεί περαιτέρω το Συμβούλιο. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με τις πέντε προτάσεις τη για τον τρόπο με τον οποίο θα προσδιοριστεί το πεδίο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τη Ελίσσα να κάνει ε, μια πιο συγκεκριμένη ε, πρόταση, γιατί είναι ακόμα πολύ ασαφή όλα αυτά, δηλαδή γενικά καταπολέμηση της, ε, του κυβερνοεγκλήματος ε, και εξασφάλιση κυβερνοασφάλειας ως καθήκοντα της υπηρεσίας αυτής. Και θα ήθελα να πω ότι αν έχουμε την πολυτέλεια να θεσπίζουμε υπηρεσίες για ένα τέτοιο και τόσο σημαντικό θέμα, καλό θα είναι να έχουμε και μια εμπεριστατωμένη εργασία που θα στηρίζει τις προτάσεις αυτές και ομολογώ εν προκειμένου ότι η επιλογή της ε, καταπολέμησης της κυβερνοεγκληματικότητας ή της, διατάραξη της διατάραξης λειτουργίας των δικτύων είναι, πιστεύω, ένα από τα ε, καθήκοντα τα οποία θα ήταν καλό να αναλάβει η ΕΝΗΣΑ και ευφυές επίσης, όπως άλλωστε έχει πει και η Επιτροπή Βιομηχανίας. Χωρίς να χρειάζεται να θεσπιστεί μια επιπλέον ε, υπηρεσία ή μονάδα κυβερνοάμυνας. Δεδομένου ότι το έγκλημα δεν γνωρίζει και οι επιθέσεις δεν γνωρίζουν σύνορα, και εφόσον θέλουμε να θεσπίσουμε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία καλό θα είναι να τις θέσουμε στη διάθεσή της τον εξοπλισμό εκείνων ο οποίος θα της επιτρέπει να καταπολεμήσει και αυτά τα φαινόμενα. Θέλει δηλαδή να έχει ένα ως το δυνατόν ευρύτατο ε, πεδίο μια ευρύτατη εντολή η ΕΝΙΣΑ και την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δυνατότητα ανάλυσης των κινδύνων, ε, των σεναρίων διακινδύνευσης, των υποδομών, των ικανοτήτων του κάθε συστήματος μέσα σε κάθε κράτος μέλος. Είναι κοινό της ε, πάση. ότι οι κρατικοί ε, υπολογιστέ, οι υπολογιστέ δηλαδή των κρατικών δομών έχουν προστασία από κυβερνοεπιθέσεις λίγο πολύ ισοδύναμη με αυτές του κάθε προσωπικού υπολογιστή που βρίσκεται σε κάθε ιδιωτικό νοικοκυριό. Άρα ανεπαρκή προφανώς και εκεί πέρα ίσω θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο ε, επίπεδο. Ε, είχαμε πρόσφατα μια επίθεση με κλοπή αντιγράφων 33 εκατομμυρίων αξίας ε, πιστοποιητικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, που πιστεύω ναι μεν ανακτήθηκαν μετά αλλά αποτελούν ένα πολύ σημαντικό σήμα κινδύνου για μας δηλαδή μας επισημαίνουν τι θα πρέπει να ε, προβλέψουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε για να αποτρέψουμε στο μέλλον τέτοιου είδους επιθέσεις τέτοιου είδου ε, επιθέσει φυσικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε στο μέλλον να εκδηλωθούν, αλλά πρέπει να είμαστε δυνατόν πιο καλά ε, προστατευμένοι απέναντί του. Αυτή τη δουλειά μπορεί να την αναλάβει η Ενίσα. Θα ήθελα όμως μια ε, οργάνωση και εντολή που θα στρέφεται προς το μέλλον, που θα έχει μακροπρόθεσμη, δηλαδή ε, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και επίσης τη δυνατότητα τόσο της φυσικής, της υλικής προστασίας, αλλά και της, ε, του ελέγχου του τρόπου με τον οποίο γίνεται η κατεργασία των δεδομένων από την ΕΝΗΣΑ, δηλαδή η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Άρα χρειάζεται η δυνατότητα της ε, παρακολούθησης των λεγόμενων data breaches, δηλαδή της ε, ε, επίθεσης ή της προσβολής ε, προσωπικών δεδομένων, αυτό τον συντονιστικό ρόλο θα μπορούσε να τον αναλάβει εμείς, αλλά θα ήθελα να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα το πράττει αυτό, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε, όπως είπα, με παραβίαση τη βασική αρχή τη προστασία των προσωπικών δεδομένων ή ευαίσθητων δεδομένων. Έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη προστασία για τον ιδιώτη από ότι από, μια κατακαιρματισμένη, ενδεχομένω ε, από ένα κατακαιρματισμένο σύστημα. Και καλύτερη ενημέρωση των εμπλεκομένων. Και όπως είπα, ε, θα πρέπει η ενίσα να είναι σε θέση να δρά προορατικά όπως λέμε. Δηλαδή να προλαμβάνει τις εξελίξεις και να αναλαμβάνει μέτρα προληπτικά. Το ίδιο μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει λίγο πολύ στο ΝΑΤΟ, ε, με τις δομές ε, του ΝΑΤΟ όπως το Cyber Security Center στο Ταλίν, στο οποίο συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου θα πρέπει, έχοντας υπόψη να αντίστοιχες δομές, να αποφεύγουμε την επικάλυψη καθηκόντων και εντολών. Να έχουμε δηλαδή στο δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και βέβαια συνεργασία μεταξύ αυτών των συγγενικών δομών. Ξέρω σε σχέση με τη Γερμανία και την αντίστοιχη υπηρεσία για την ε, προστασία από το κυβερνοέγκλημα ότι υπάρχουν κάποιες γενικές ιδέες που προβάλλονται ως ε, στόχοι για το έργο και την αντολή που θα πρέπει να αναλάβει αυτή η αποκεντρωμένη υπηρεσία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσω τώρα, μάλλον θα πρέπει να έρθει ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή, εκτό και αν θέλετε να συνεχίσω, γιατί πάντα θα βρίσκω κάτι να ε, πω στην υπόθεση αυτή, αλλά μάλλον δεν θα με παρακολουθείτε πια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το πνεύμα συνεργασία που δείξατε, κύριε Αλβαρό ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ε, ήταν, ε, ήρθε μόλις αρχίσατε να μιλάτε. Οπότε δεν χρειάζεται να συνεχίσετε. Θα ακούσουμε την εξήγηση της προτάσης της Κομισιόν από την ίδια την Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο. Ε, είχα όμως έτσι την ευκαιρία να ακούσω τον κύριο Άλβαρο. Οπότε στην παρουσίασή μου θα θα σχολιάσω και ορισμένες από τις δικές του παρατηρήσεις. Θα σας παρουσιάσω την ε, πρόταση κανονισμού για τον ΕΝΙΣΑ. Ε, υπήρχε ήδη αυτή η πρόταση στην ε, ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη ως δράση κλειδί υπαριθμών 6 για την ενίσχυση ενός ψηλού επίπεδου πολιτικής δικτύων ε, συμπεριλαμβανομένης και, και, της, ε, και του εξυγχρονισμού της, ε, του οργανισμού ΕΝΙΣΑ. Έλαβαν, έλαβε χώρα δημόσια διαβούλευση και για την ΕΝΙΣΑ και για, την, για το θέμα των εργαλείων ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτές οι διαβουλεύσεις έγιναν από το 2007 στο 2009. Επίσης, εκδόθηκε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου για την... Ε, ε, μάλλον το Δεκέμβριο του 2009 για την προσέγγιση, συνεργατική προσέγγιση σε ό,τι αφορά το θέμα, τα, θέμα ασφάλειας ε, δικτύων και πληροφοριών. και εξετάσαμε πέντε εναλλακτικές λύσεις. Πρώτον, μηδενική πολιτική, χωρίς επέκταση της εντολής στην ενίσα. Δεύτερον, ε, συνέχιση της εντολής, απέκτα, ε, παράτασή της ε, με τους ίδιους όρους με τους σημερινούς τρίτων, διεύρυνση των λειτουργιών του οργανισμού για να λάβουμε υπόψη εξελίξεις στο θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Εκεί έχουμε γρήγορες εξέλιξεις πράγματι. Τέταρτον, να δώσουμε στην, στον οργανισμό επιχειρησιακές αρμοδιότητες για την καταπολέμηση των εγκλημάτων του κυβερνοχώρου. Ε, ε, ε, η τιμή, το κόστος όμως μιας τέτοιας διεύρυνσης θα ήθελα να σας ότι είναι πολύ ψηλό. Θα απαιτούσε διαφορετικές πολιτικές από τις σημερινές που ασκούνται στον οργανισμό. Ο προπολογισμό του οργανισμού θα έπρεπε να τετραπλασιαστεί τουλάχιστον. Και πέμπτη, πέμπτο σενάριο, η, πάνω πέρα από, το, από την τέταρτη εναλλακτική λύση, ε, να δώσουμε στην, ε, στον οργανισμό ε, και τα μέτρα, τα μέσα, τα απαραίτητα μέσα για την καταπολέμηση του, του, του εγκλήματος στον κυβέρνο χώρο. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την σημερινή εντολή της ΕΝΗΣΑ. Η ΕΝΗΣΑ στην η Κομισιόν στην πρότασή της έχει αυξήσει την ε, ευελιξία της, ε, του οργανισμού, ε, τα καθήκοντα του οργανισμού την χάνουν μια πιο γενικής περιγραφής, έτσι ώστε να μπορεί ο οργανισμός να αντιμετωπίσει και μελλοντικές προκλήσεις, οποίες αγνοούμε αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά η περιγραφή αυτού των καθηκόντων είναι αρκετά σαφή έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι όπω σα είπα. Δεύτερον, μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με την ε, κανονιστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή όλα τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μπορούν να προσφεύγουν στον, στην ενίσα προκειμένου να λαμβάνουν συμβουλέ. αυτό ευθυγραμμίζεται με τι κανονιστικέ κανονιστικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, η εντολή προτείνουμε ε, καθιστά την ενίσα ενδιάμεσο ανάμεσα στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών και στην καταπολέμηση του, των εγκλημάτων του κυβερνοχώρου. Ο οργανισμός δεν λαμβάνει αρμοδιότητες για καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, αλλά θα αποτελεί γέφυρα έτσι ώστε οι, ε, οι φορείς που ασχολούνται με την καταπολέμηση του εγκλημάτου του κυβερνοχώρου θα γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται στο θέμα της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών και αντιστρόφως. Η πρότασή μας ε, έχει με αυτόν τον τρόπο στόχο να προσθέσουν τις, τους φορείς προστασίας δεδομένων και ε, επιβολής του νόμου στους ε, φορείς που συνεργάζονται με την ΕΝΗΣΑ. Ε, μετά, ένα σημαντικός εποπτικός ρόλος δίνεται στο, ε, εκτελεστικό ε, συμβούλιο της, ε, στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού και δίνεται η δυνατότητα σε αυτό να εκδίδει γενικές κατευθυντήρες ραμές, δηλαδή με άλλα λόγια να καθορίσει μια μακροπρόθεσμη πολιτική. Η καθημερινή διαχείριση θα, θα παραμείνει αρμοδιότητα του εκτελεστικού διευθυντή όμως. Πέμπτον, απλοποίηση των διαδικασιών ορισμένες ε, διαδικασίες αποδείχθηκε ότι ήταν ε, υπερβολικά επαχθείς. Για παράδειγμα, στην υπάρχουσα στην ισχύουσα εντολή κάθε χρόνο η Κομισιόν ε, εκδίδει γνωμοδότηση για το προσχέδιο προγράμματος εργασίας της ΕΝΙΣΑ. Αυτό εγκρίνεται από το, την Ολομέλεια των Επιτρόπων. Ε, τώρα πια θα εγκρίνεται αυτή η γνωμοδότηση από τις υπηρεσίες της Κομισιόν χωρίς να χρειάζεται να φτάνουν στο Κολέγιο των Επιτρόπων κάθε φορά. Ε, ε, επίσης προβλέπουμε την δυνατότητα παράτασης της αιτίας του εκτελεστικού διευθυντή που ε, διορίζεται για πέντε χρόνια. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να παραταθεί για τρία έτη ή θητεία. Έβδομον, σταδιακή αύξηση του προϋπολογισμού του οργανισμού. Μας ελέγχθη ότι δεν είναι δυνατόν να ε, εξασφαλίσουμε ε, κονδύλια για όλο το χρονικό διάστημα το οποίο καλύπτει η πρότασή μας, γιατί ο προϋπολογισμός μετά το 2013 θα πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο ε, του πολιετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου. Συνεπώς όλα τα στοιχεία για μετά το 2013 λείπουν. Θα τα προσθέσει η Κομισιόν όταν γίνει σαφής, σαφές ε, το, χρηματο, το δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, το πολιετές, ε, συγγνώμη, χρηματοοικονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2013. Μετά σε ό,τι αφορά τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ασφάλειας του κυβερνοχώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην, Κομισι... και στην Κομισιόν. χρειάζεται να συντονίσουμε τι δραστηριότητε, αυτέ, τι δραστηριότητε τη ΕΝΗΣΑ και τις δραστηριότητες καταπολέμηση του εγκλήματο στον κυβερνοχώρο. Όμω, λέμε ότι όλε αυτέ οι δραστηριότητε δεν μπορούν να μπουν στην ίδια ομπρέλα ακριβώ. γιατί οι ε, εμπλεκόμενοι φορεί είναι διαφορετικοί, οι προπολογισμοί είναι διαφορετικοί και οι στόχοι είναι διαφορετικοί. Χρειάζεται να γίνει όμως συντονισμός και λαμβάνει χώρα ήδη στο εσωτερικό της Κομισιόν. Όμως δεν θα μπορούσαν αυτοί οι τρεις τομείς να ενσωματωθούν σε ένα, να ενοποιηθούν. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση της πρότασης. Έχοντας ακούσει τον εισηγητή τον κύριο Αλβάρο μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Σόνικ και κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Κύριε Σόνικ, έχετε το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση που αφορά την ενίσα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη την ανάλυση του κόστους και αποδοτικότητας. Αυτό έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσω τι σχέσει με τα άλλα κράτη-μέλη όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια. Η ΕΝΙΣΑ μόλις τώρα προσφέρει υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίως προσέφερε υπηρεσίες προς τα εμπορικά επιμελητήρια πιο αραιά μάλλον ε, προσφέρει υπηρεσίες προς τα εμπορικά επιμελητήρια και άλλους φορείς. Άρα είναι περιορισμένο το, περιορισμένη η εμβέλεια του φορέα αυτού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποστηρίζει τον πολλαπλασιασμό των φορέων στην Ευρώπη γιατί δυσκολεύεται η εξολόγηση. Θα υποστηρίξει όλες τις αλλαγές που έχουν σαν στόχο όμως την καλύτερη λειτουργία του φορέα και την κάλυψη των αναγκών. Πρέπει να εξετάσουμε τη λειτουργία αυτού του οργανισμού. Ποιοι φορεί συμπεριλαμβάνονται, ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία της ιδιωτική ζωής κλπ. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με, την, με τον οργανισμό αυτό. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει περισσότερες προκλήσεις όπως πολέμη του κυβερνοεγκλήματος. Θα πρέπει να είναι ένα κέντρο αριστείας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των δεδομένων, ηλεκτρονικών υπογραφών και γενικά την πρόθεση υψηλών προδιαγραφών όσον αφορά την πληροφορική. Για την καταπολέμηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και την αντιμετώπιση των διαφόρων απειλών και του hacking, Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, χρειάζονται περισσότερες συζητήσεις. Άλλες πτυχές, η έδρα του οργανισμού έχει σημασία, δεν είναι πολύ στατηγική η τοποθεσία, δεν είναι εύκολα προσβάσιμη. Από την άλλη γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν διάφοροι οργανισμοί να είναι στην επικράτειά τους. Όσον αφορά το Γενικό Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο, Αυτά πρέπει να λυθούν με διαφάνεια. Θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια. Η Πολωνική Προεδρία θα αναλάβει αυτά τα θέματα, θα πραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ μέρου του Συμβουλίου σχετικά με τον ε, κανονισμό. Και αυτά είναι όλα όσα είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. παπα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Αλβάρο, τον εισηγητή μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και την πολύ σημαντική συζήτηση. Χρειαζόμαστε την ΕΝΙΖΑ, πράγματι. Όταν δημιουργήθηκε το 2004 η ΕΝΙΖΑ, δεν γνωρίζαμε πιθανότατα το στεγγής μέλλον οι προκλήσεις θα αυξανόταν. Το 2011 οι προκλήσεις πράγματι είναι πολύ μεγάλες ο ρόλος της ΕΝΙΖΑ μπορεί να είναι κρίσιμη σημασία. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Αναφέρομαι στο ψηφιακό πρόγραμμα, στο κυβέρνο έγκλημα. Συζητήσαμε πριν τις εμπιστευτικές πληροφορίες, τις σημαντικές πληροφορίες. Όλα αυτά είναι κρισίμου σημασίας. Η ΕΝΙΖΑ βέβαια πρέπει να είναι σημαντικός θεσμός που θα διδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την έδρα της. Χαίρομαι ότι δεν συζητήσαμε εκτενώς το θέμα σε αυτή την Επιτροπή. Στην Επιτροπή ίντε διεξήχθη. Έγινε μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ένα σχόλιο έχω μόνο πάνω σε αυτό. Το νησί της Κρήτης είναι το μεγαλύτερο ελληνικό νησί. Ο κ. Αλβάρο είπε ότι είναι καλό μέρος για να διασκεδάζει κανείς. Να επενθυμίσω στους συναδέλφους ότι εκατοντάδες χιλιάδες ε, πληθυσμό έχει Κρήτη. Ζει ο κόσμος εκεί, εργάζεται, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έχουμε έξοχες υποδομές στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, δικτύωση και τα συναφή ζητήματα. Βεβαίως δεν έχουμε μόνο τα νησιά που αποτελούν μια χώρα, έχουμε και νησιά που είναι αυτά κάθε αυτά χώρες, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Μάλτα. Δεν πιστεύω ότι επειδή η Κρήτη είναι νησί, αυτό σημαίνει ότι είναι κακό μέρος για να εδρεύει, να είναι εκεί η Ενίζα. Έχω επιστολές, ανακοινώσεις ελληνικής κυβερνήσεως σχετικά με την τοποθεσία, σχετικά με την Κρήτη, ότι είναι καλή επιλογή για μας. Εν πάση περιπτώσει, αν χρειαστεί οι συνάδελφοί μας να έχουν περισσότερες πληροφορίες, είμαι στη διάθεσή τους, έχω μαζέψει πολλές πληροφορίες, οπότε αν χρειάζεστε κάτι σας παρακαλώ να μου το πείτε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Άλμπρεχτ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Άλβαρο, για τη δουλειά του. Δεν έχω πολλά να προσθέσω προς το παρόν. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ, διότι επανέρχεται συχνά και έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες αυτές της υπηρεσίας. Είναι πολύ σημαντικό να τη συζητήσουμε, διότι δεν αποτελούν αυτό σκοπό της υπηρεσίας. Η δραστήρια αντιμετώπιση της κυβερνοεγκληματικότητας ή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η υπηρεσία αυτή έχει θεσπιστεί για να εξασφαλίσει την τεχνολογική ασφάλεια της ε, διακίνησης πληροφοριών. Και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να περιοριστούμε. Εάν αρχίσουμε να συζητούμε το πώς θα διευρύνουμε το πεδίο δραστηριοτήτων αυτής της υπηρεσίας, θα φτάσουμε μέχρι και το πρόβλημα που συζητούσαμε νωρίτερα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, των εκτελεστικών δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων τέτοιου είδους υπηρεσιών, των κανόνων που ισχύουν για τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών και πολλών άλλων ζητημάτων τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ε, εν λόγω διεύρυνση αρμοδιότητων. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω θα πρέπει να περιοριστούμε στην τεχνολογική ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών. Αυτό είναι όλο. Σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε, αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε, να αναπτύξουμε. Αυτό είναι ο στόχο τον οποίο επιδιώκουμε στη τελευταία ανάλυση. Και τώρα ο κ. Αλβάρο θα μα ξαναπεί κάτι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ας αρχίσω από το τέλος. Με ναι, γνωρίζω, κύριε κύριο αρκετά καλά. Ώστε να ξέρω ότι δεν σκοπεύω να θεσπίσω NSA, μυστική υπηρεσία πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας καλύτερα αλλά πρέπει να δούμε και σε πόσο βαθμό, σε ποιο βαθμό ξέρουμε τι κάνει η ΕΝΕΣΑ. Δηλαδή, μια υπηρεσία η οποία έχει αυτόν τον τεχνολογικό έλεγχο της ασφάλειας πρέπει να είναι και σε θέση να αποστείλει ένα σήμα κινδύνου. Ένα ιός μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να ε, μολύνει δίκτυα ολόκληρα. Έχουμε δει στη σήμερον ημέρα τα μεγέθη της ζημιάς που μπορεί να αγγίξει η ε, διάδοση ενός ιού μέσα από τα συστήματα. Ε, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για δημόσιους οργανισμούς, οποιοδήποτε εντό αγωγικών πελάτης ε, θα αναγνωρίζει ασφαλώς τη σημασία της real-time καταπολέμησης, καταπολέμησης, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο των επιθέσεων τέτοιου τύπου από την ΕΝΙΣΑ και πιστεύω ότι μπορεί να το προσφέρει αυτό η ΕΝΙΣΑ, δηλαδή την επιτήρηση της ασφάλειας και όχι μόνο την τεχνολογική ε, διασφάλιση. Αυτό είναι το ένα. Ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο φυσικά μπορούμε με την άνεσή μας να συζητήσουμε, δεν έχω καμιά αντίρρηση, αλλά πρέπει και να έχουμε υπόψη ότι εάν αναγνωρίσουμε ε, και σε άλλου τομεί, όπω φέρει πίνη στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπου εγώ είμαι ο πρώτο που αγωνίζεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. να γνωρίσουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν μόνο εδαφικέ πτυχέ αυτών ε, των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα και τη ε, υπερσυνοριακή προστασία του, τότε χρειαζόμαστε και ένα σύστημα προστασία προσωπικών δεδομένων από ενδεχόμενες επιθέσεις μέσα από τα δίκτυα που θα καλύπτει ολόκληρη την επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωση και ενδεχομένω θα έχει και συνεργατική δράση με άλλες αντίστοιχε υπηρεσίες όπως είπα νωρίτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια καλή πρόταση αλλά δεν είναι επαρκή, δεν ήταν αρκετά θαραλέα η πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ περαιτέρω στι διεκδικήσει τη για την ενίσχυση, για τα καθήκοντα που θα μπορούσε να λάβει αυτή. Θα πρέπει να δούμε και πόσα χρήματα, με λίγα χρήματα προφανώ δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα η, ε, εάν έχει μόνο μια ε, συμβουλευτική δραστηριότητα προφανώς δεν λύνει πολλά προβλήματα και αν δεν λύνει πολλά προβλήματα μάλλον και τα λίγα χρήματα που κοστίζει είναι πεταμένα από το παράθυρο. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να προβλέψουμε μια κατάλληλη, ε, μια κατάλληλη χρηματοδότηση. Και ε, για καλή του στίχη είμαι και συντάξει από την Επιτροπή των Προϋπολογισμών για αυτά τα θέματα και άρα θα το κοιτάξω και από αυτή την πτυχή. Βέβαια, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη το δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν είμαστε σίγουροι για, τα, ε, για τον πολιετή σχεδιασμό, τι είδου ε, κονδύλια θα μπορούσαμε να διαθέσουμε ε, για την υπηρεσία αυτή, όπω και για τι άλλε. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω τώρα ένα ζήτημα σχετικό με τις ε, προσβολές όπως αυτή την ιστορία με τα 33 εκατομμύρια ευρώ αξίας των πιστοποιητικών για τις εκπομπές ευρωπαϊκών πιστοποιητικών για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα πόσο μεγάλος ήταν ο κίνδυνος και πόσο συγκεκριμένα επιθέσεις οι οποίες στοχεύουν είτε πρόκειται για τράπεζες, είτε πρόκειται για δημόσιους οργανισμούς, ε, είτε πρόκειται για αντίστοιχους μεγάλους φορείς, οι επιθέσεις αυτές μπορούν να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Και αυτή η αυτές οι επιθέσεις θα πρέπει να δυνατόν να αντιμετωπιστούν από μια υπηρεσία τέτοια, η οποία, ναι, θα πρέπει, πιστεύω, να ε, υπάγεται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και όχι να ε, διακλαδώνεται και να μεγενθύνεται κατά τρόπο ανεξέλεγκτο και να ξεφεύγει του ελέγχου μας. Αυτό άλλωστε επεσήμαναν και άλλοι συνάδελφοι. Και ξέρω και φαντάζομαι ότι το ίδιο θα σημαίνευε και αν ήταν η ε, δική μου η πατρίδα, τον Τίσσελντορφ, η έδρα τη υπηρεσία, ότι ο κύριο με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και πάθο υποστηρίζει την έδρα τη Κρήτη για την ε, υπηρεσία αυτή. Ο Σάιμον ε, πιστεύω δεν θα με παρεξηγήσει εάν ε, πω ότι θα μπορούσε εξίσου η Μάλτα ή η Κύπρος να είναι η έδρα της Υπηρεσία αυτή και να εντόπιζα αντίστοιχα προβλήματα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με την ανάγκη, κατά την έποψή μου, να υπάρχει ένα μεγάλο αστικό κέντρο, ένα κέντρο το οποίο θα στηρίζει τις λοιπές δραστηριότητες υπηρεσίας αυτής και παρακαλώ να μην θεωρήσουν οι συνάδελφοι, ε, τα λόγια μου θεωρώ ότι είναι εξαίρετη η ιδέα της έδρας μιας της υπηρεσίας σε ένα νησί, δεν αποτελεί εμπόδιο νησιωτικό χαρακτήρας, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ίσως θα έπρεπε να δούμε και το σε ποιο βαθμό υπάρχει ε, δυνατότητα για ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων αυτή τη υπηρεσία. Δεν έχω καμία πρόθεση, επουδενή την πρόθεση, να αρνηθώ στην Ελλάδα ω κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να υποδέχεται μια τέτοια υπηρεσία στην επικράτειά τη. Απλώ θα πρέπει ίσω να ενισχυθεί η λειτουργία τη κατά κάποιο τρόπο. Ε, άλλες δραστηριότητες λοιπόν, όπω είπαμε, κονδύλια επιπλέον, όπω είπαμε επίση, για την ενίσα και όπω είπα Ανησυχώ βαθύτατα για το γεγονό ότι ενδεχομένω, αφού έχουμε περάσει όλη αυτή τη συζήτηση και έχουμε ε, δαπανίσει τόσο χρόνο να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, μπορεί τελικά να ε, συρρυκνωθεί σε ένα μόνο τεχνολογικού χαρακτήρα ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Έχει κάποια σχόλια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά αυτή την παρουσίαση, θέλει να πει κάτι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παρακολούθησα τη συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα πράγμα που θέλω να διευκρινίσω ή μάλλον να διαλύσω μια παρεξήγηση. Υπόθηκε σε κάποια φάση ότι η ενίσα δραστηριοποιείται τώρα βασικά παρέχει υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν ισχύει. Η ΕΝΙΖΑ δραστηριοποιείται όλος ιδιαίτερος ε, με διάφορους ε, εμπλεκομένους φορείς, παρέχει υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, καλύπτει ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διεξάγονται συζητήσεις και με τους δύο τομείς, οπότε αυτό είναι αναγκαίο. Και εάν έπρεπε να καθορίσουμε πού είναι το κέντρο βάρους των παρεχομένων υπηρεσιών της ΕΝΙΖΑ, θα έλεγα ότι είναι προς τα κράτη-μέλη περισσότερο, παρά προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την ώρα. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you. Now, now Νομίζω ότι κλείνουμε με αυτό το σημείο. Όπως σας είπα, η κυρία Μάλστρομ θα φτάσει γύρω στις 12.30. Θα συναντηθεί με τους συντονιστές, οπότε προτείνω να κηρύξουμε την λήξη της, ε, της συνάντησής μας μέχρι τις 3. Θα ξανασυναντηθούμε στις 3 το απόγευμα μετά τη συνάντηση των συντονιστών και αφού Εκεί ακούσουμε την Επίτροπο Μάλστρομ. Ευχαριστώ.